σχέση με τα βασανιστήρια από τη CIA. Πρώτος ως εκπρόσωπος ε, του Συμβουλίου θα λάβει τον λόγο ο Υπουργός Ντελαβέντοβα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί κύριοι βουλευτές. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ένα εταίρο σημαντικό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Όμω, Υπήρξαν κάποιες σοβαρές ανησυχίες και διαφορές μεταξύ ημών για διάφορα στοιχεία της πολιτικής κατά της τρομοκρατίας που ασκεί η ΕΠΑ. Εμείς ξεκινήσαμε το διάλογο με τις, Ηνωμένε με επί χρόνια και σήμερα θα συζητήσουμε για μια έκθεση της Γερουσίας που αφορά ένα παλιό αμερικανικό πρόγραμμα που έχει ολοκληρωθεί επισήμως πια εδώ και έξι χρόνια. Συμμεριζόμαστε την άποψη που εκφράστηκε από τον πρόεδρο Ομπάμα, με βάση την οποίο αυτές οι τεχνικές είναι αντίθετες σε αυτές τις αξίες που υπερασπιζόμαστε και δεν είναι χρήσιμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε αυτή τα, αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό χαιρόμαστε για τη δημοσίευση αυτής της έκθεση για να ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση. Αυτό δείχνει το άνοιγμα και τη διαφάνεια και την διάθεση να αναγνωριστούν τα παλιά λάθη. Το Συμβούλιο έχει πει κατ' επανάληψη ότι ο αγώνας κατά της τρομοκρατία θα πρέπει να γίνει με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να σεβαστούμε το ύψιστο διεθνές δικαίωμα, το ανθρωπιστικό δικαίωμα καθώς και το δικαίωμα των προσφύγων. Σε ό,τι αφορά ε, τα δικαιώματα αυτά, αυτά αποτελούν βασικό στοιχείο τη στρατηγική κατά τη τρομοκρατία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κέντρα αυτά κράτησης που δημιούργησε η CIA ε, αποκαλύφθηκαν το 2006 και τότε είχαμε πει ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι στην, ε, στο βασανιστήρια και σε απάνθρωπες ε, συμπεριφορές. Από την έκθεση της Γερουσίας προκύπτει ότι Εγκρίθηκαν διάφορες τεχνικές ε, όπως αυτές που προαναφέραμε. Από το 2006 η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε ένα τακτικό ε, διάλογο με τους Αμερικανούς ομολόγους για τα θέματα, τα νομικά στοιχεία της, ε, του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Και έχουμε υποβάλει στις ΗΠΑ μια σειρά από ερωτήσεις και ανησυχίες. Επιμείναμε δε στην ανάγκη να σεβαστούμε το διεθνές δικαίωμα και τα ανθρώπινα δικαιώματα το διεθνές δίκαιο, συγγνώμη. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι ο πρόεδρος Ομπάμα ολοκλήρωσε επίσημα το πρόγραμμα της ΣΥΑ, το τερμάτισε δηλαδή, λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Και με διάταγμα είχε απαγορεύσει κάθε βασανιστήριο και κάθε έντονη τεχνική ανάκρισης όπως λεγόταν. Είχε ζητήσει επίσης να μην διαχειρίζεται η CIA τα κέντρα αυτά και είχε απαγορεύσει τις, τεχνικές, ε, τις έντονες τεχνικές ανάκρισης. Μετά από μια κοινή δήλωση τον Ιούνιο του 2009, εμείς με τις Ηνωμένες είχαμε πει ότι θέλουμε να επανεξετάσουμε αυτές τις πολιτικές σε ό,τι αφορά την κράτηση, την μεταφορά, τις ανακρίσεις που χρησιμοποιούμε για την ε, καταπολέμηση τη δημοκρατίας και θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαφάνεια στις πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν στα πλαίσια αυτών των πολιτικών. Ε, όπως επίσης θα πρέπει, είχαμε πει ότι θα πρέπει να καταργηθούν και τα μυστικά κέντρα κράτησης. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία μόνο αν πιστεύουμε στις αξίες μας, τις θεμελιώδεις μας αξίες. Η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου μπορεί να οδηγήσουν από μόνες τους σε τέτοια μνησικακία και να οδηγήσουν από μόνε τους στην προσφυγή, στην τρομοκρατία. Και επίσης δεν δικαιολογούνται ποτέ. Αυτές οι πολιτικές, παρότι υποτίθεται πολεμού την τρομοκρατία, μπορούν να δημιουργήσουν τις κατάλληλε συνθήκες για να διαδοθεί η τρομοκρατία. Επί χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιορίστηκε στην έναρξη διαλόγου με τι ΗΠΑ, αλλά προώθησε και συγκεκριμένε δράσει για να προωθήσει αλλαγέ στην Αμερικανική πολιτική. Φερρυπίν το 2009 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα πλαίσιο που διευκόλυνε την ε, υποδοχή από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρώην κρατουμένο στον Κουαντάναμο υποστηρίζοντας τον ε, στόχο του Προέδρου Ομπάμα να κλείσει τον Κουαντάναμο μέσα σε ένα χρόνο. Έγινε επίσης μια ενδελεχής ε, αναθεώρηση των Αμερικανικών πολιτικών κατά της δημοκρατίας με βάση το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα περιμένοντας μία αρρύθμιση των σχετικών πολιτικών προβλημάτων. Τώρα στο Αφγανιστάν, στη Συρία και στο Ιράκ, ε, στους αγώνες αυτούς, πολέμους αυτούς, είχαμε σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία μία προσέγγιση που βασιζόταν στην δημοκρατία. Οι ένοχοι θα πρέπει να διωχθούν με βάση τις αρχές του ποινικού δικαίου έχουμε μακρά εμπειρία σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των τρομοκρατών. Οι έρευνες των κατασταλτικών αρχών είναι σημαντικές για να πάρουμε πληροφορίες για τρομοκρατικά δίκτυα και για να ακυρώσουμε τις προθέσεις τους. Και χάρη στις προσπάθειες αυτές ε, βάλαμε εκατοντάδες τρομοκράτες ε, πίσω από τα σίδερα. Θεωρούμε ότι η εθνική ασφάλεια είναι αρμοδιότητα κάθε κράτους μέλους. Αυτό σημαίνει ότι η δουλειά της υπηρεσίας πληροφοριών των Ε.Π.Α. εκφεύγει της ε, αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμικών της οργάνων. Και οι έρευνες για την εμπλοκή των ΗΠΑ στα προγράμματα της CIA είναι αρμοδιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών και ουχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατα... Κατακλείδη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευμένα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δράσεις που προωθήθηκαν για να καταπολεμήσουν τον... τη δημοκρατία ελέγχονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου. Πέρα, επίσης, πέρα, μετά την θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας, ε, μπορούμε να επανεξετάσουμε την ε, νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την εσωτερική ασφάλεια. Θα πρέπει να έχουμε ένα κατάλληλο πλαίσιο στο εσωτερικό του οποίου μπορούμε και οφείλουμε να καταπολεμήσουμε τη μάστιγα της τρομοκρατίας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη δήλωση του Συμβουλίου. Τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής, ο Επίτροπος κ. Σαβραμόπουλος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την οποία εκπροσωπώ απόψε εδώ για αυτό το θέμα, είναι όπως και εσείς <clears throat> φρικιά για αυτά τα ευρήματα όσον αφορά την έκθεση της ε, Γερουσίας για τόσα έκανε η CIA Μέρος από αυτά αποκαλύφθηκαν για την 9η Δεκεμβρίου. Όπως γνωρίζετε το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ε, ερευνητικών διαδικασιών είναι διαβαθμισμένο. Αυτή η έκθεση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα όσον αφορά σοβαρές παραβιάσεις ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων από τις αρχές των ΗΠΑ και άλλων ατόμων που υπηρετούν τη CIA, CIA μεταξύ 2001 μέχρι τον Ιανουάριο 2009. Όπως και ο πρόεδρος Ομπάμα εξάλλου πολύ σωστά είπε κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, οι πράξεις, οι ενέργειες αυτές υπό το πρόγραμμα της CIA αντέβαιναν τις αξίες των ΗΠΑ, αναγνωρίζοντας έτσι ότι ένα από τα πιο αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι να παραμείνει κανείς πιστός στις αρχές και τις αξίες και τα ιδανικά των ΗΠΑ που εκπροσωπούν οι ΙΠΑ. Και αυτό είναι εκείνο το οποίο τον οδήγησε το, κατά τη διάρκεια του έτους 2009 <clears throat> χωρίς καμιά αμφιβολία να καταδικάσει τα βασανιστήρια, κάτι το οποίο χειροκροτήσαμε τότε εμείς. Και αυτό επειδή αυτό είναι η πραγματική ουσία όσον αφορά τα βασανιστήρια. Είναι όχι μόνο λάθος, είναι έγκλημα τα βασανιστήρια. Είναι μια εγκληματική πράξη και ποτέ δεν πρέπει να, να γίνονται βασανιστήρια. Και ενώ είναι ανησυχητικά αυτά τα ευρήματα της ε, Επιτροπής της Γερουσίας, ε, δεν είναι μια ε, απόλυτη έκπληξη διότι οι πτήσεις, μυστικές πτήσεις παράδοσης κρατουμένων και η κακή μεταχείριση των κρατουμένων από την CIA μέσα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας από την ΗΠΑ ήταν κάτι που μας ανησυχούσε ιδιαίτερα από τότε που δημοσιεύθηκαν αυτά πριν από 10 χρόνια περίπου. Και από τότε, έκτοτε, αρκετά τι φορείς και σώματα των Ηνωμένων Εθνών, Ειδική ειδικοί ε, επίτροποι και ε, καθώς επίσης και το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασαν εξίσου όλοι αυτές τις πρακτικές που τώρα τεκμηριώνονται από αυτή την ε, έκθεση της Επιτροπής της Γερουσίας. Αυτό το σώμα είχε εμπλακεί σε αυτή τη διαδικασία ευθύ εξ αρχής... με την απόφαση να συσταθεί, να συγκροτηθεί μια επιτροπή ώστε να υπάρξουν και δύο εκθέσει ιδία πρωτοβουλία κατά το 2007 και το 2012 ε, εξίσου, καταδικάζοντα αυτές τις πρακτικές και εκφράζοντας ε, την ανάγκη να υπάρξει, να προαχθούν και να προστατευτούν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και όπως ε, και από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτά τα θέματα τα θίξαμε, τα αναφέραμε σε σχέση με τη ΣΥΠΑ με αρκετές ε, αφορμές, με επιστολές από την Προεδρία του Συμβουλίου και στον κανονικό τακτό διάλογό μας όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τον σεβασμό των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι ένα θετικό βήμα αυτή η έκθεση της Επιτροπής Γερουσίας ώστε δημόσια να αντιμετωπιστεί ο τρόπος με τον οποίο οι ευθύνε αυτές της CIA όσον αφορά τη διεξαγωγή ε, βασανιστήριων και την κακομεταχείριση αυτών που βρισκόντουσαν ως κρατούμενοι στην, ε, ε, υπό την εξουσία των Αμερικανικών αρχών. Πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αποσαφινιστούν απόλυτα αυτά τα συμβάντα σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, συμπεριλαμβάνοντας επίσης και τις ατομικές ευθύνες που πρέπει να διακριβωθούν για εκείνους που ενεπλάκησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει κάθε μορφή βασανιστήριων και κακομεταχείρισης υπό οποιασδήποτε συνθήκες και πρέπει <clears throat> σε σχέση με την εκρίζωση και αντιμετώπιση κάθε μορφής τέτοιας πρακτικής στην Ευρωπαϊκή, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια να καταβάλουμε προσπάθειες ως προτεραιότητα της πολιτικής μας ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως επανειλημμένα έχει υπογραμμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσπάθειες ε, που γίνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να διεξάγονται με έναν τρόπο που θα ανταποκρίνεται και θα συνάδει με τους κανόνες δικαίου και θα σέβεται τις κοινέ μας αρχές και αξίες θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις μας ε, υπό το διεθνές δίκαιο όπως απορρέουν αυτές. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις αρχές για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, για τους πρόσφυγες και την ανθρωπιστική ε, συνιστόσα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε τονίσει ευθύ εξ αρχή ότι όλα τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να διεξαγάγουν σε βάθος ανεξάρτητες αναλύσεις και αμερόληπτες ε, ε, εξεταστικές ενέργειες ώστε να διακριβωθεί το τι ακριβώς συνέβη σε σχέση με τη CIA. Πρέπει να αποσαφινιστούν οι ευθύνε και να μπορέσουν τα θύματα να αποζημιωθούν για τα όσα υπέστησαν. Αυτό υπενθυμίστηκε σε μια κοινή επιστολή που απεστάλησε όλα τα κράτη-μέλη το 2013. Από τον, την τότε αντιπρόεδρο Ρέντινγκ ε, και την επίτροπο Μάλστρομ. Γνωρίζουμε ότι οι αρχές των κρατών μελών, δικαστικές αρχές των κρατών μελών έχουν κατά το παρελθόν αναλάβει πρωτοβουλίες ε, διακριβωτικές όσον αφορά πράκτορες της CIA, όσον αφορά την απαγωγή, σύλληψη, μεταφορά, παράνομη κράτηση, βασανιστήρια και κακομεταχείριση υπόπτων υπό ε, το πρόγραμμα ε, φυλάκισης υπόπτων της CIA. Την ίδια ημέρα όπως δημοσιοποιήθηκε αυτή η ε, έκθεση μάθαμε από τον τύπο ότι το κέντρο ε, κράτησης ε, στο ε, Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν δύο από τους κρατούμενους που είχαν παραδοθεί στις αρχές βρισκόντουσαν υπό την υποκράτηση από το 2002 ακόμα και αρκετά χρόνια υπό την υποκράτηση της CIA χωρίς να έχει διεξαχθεί δίκη. 106 κρατούμενοι παραμένουν ακόμα στο, στη φυλακή Γουαντάναμο καθώς και κρατούμενοι που δεν έχουν ούτε προσαχθεί σε δίκη, ούτε έχουν αθωωθεί ώστε να αφαιθούν ελεύθεροι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθήσει εκ του σύνεγγυς να παρακολουθεί αυτή την κατάσταση και θα αναφέρει πάντα τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας με τις ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτρεπε. Θα ακούσουμε τώρα τους ομιλητές εξ των πολιτικών ομάδων. Η Μόνικα Χολμάιερ για δύο λεπτά από πλευρά ΤΕΛΚ. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Προεδρία του Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση που μέσω της Επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ κατατέθηκε είναι μια πολύ ανησυχητική έκθεση. Όταν λέει ο πρόεδρος Ομπάμα ότι δείχνει την φρίκη των δράσεων της CIA παγκόσμια και υπονομεύεται έτσι η αξιοπιστία και το κύριο στον είπα 100% συμφωνώ μαζί του. Πρόκειται για το ζήτημα ουσίας είναι μπορούμε να προστατέψουμε τα ιδανικά μας ε, όταν ποδοπατούμε τις αξίες και τις αρχές μας ε, κατάφορα. Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί υπό το πρίσμα του ΕΛΚ. Και εγώ προσωπικά απαντώ όχι. Δεν μπορούμε αυτά τα ιδανικά, αυτές τις αρχές και αξίες να τις ποδοπατούμε. Όποιος ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα, <clears throat> τα δικαιώματα του ανθρώπου και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου δεν μπορούν να θίγονται και να παραβιάζονται είναι απαραβίαστα. Αλλά για την κάθε μέθοδος όπως η τρομοκρατία και οι πιο ε, ακραίες μέθοδοι ανακρίσεων δεν ανήκουν στους καταλόγους εκείνους που θεωρούνται μέσα αποδεκτά. Το waterboarding όπως ε, το ανέφερε και ο κύριος Μακέιν υπό, το, υπό την δική του άποψη και ιδιαίτερα αξιόπιστη όπως τα περιέγραψε είπε ότι οι Αμερικανοί με αυτή τη μέθοδο με το waterboarding επί πολλά χρόνια είχε, είχαν ασκήσει αυτή τη μέθοδο. Αυτό, αυτό το οποίο κατηγορώντας άλλους ε, που άσκησαν αυτή τη μέθοδο δεν μπορούν οι ίδιοι να την ακολουθούν. Και σε σχέση με την αμερικανική κοινοβουλευτική παράδοση αυτό τούτου είδους ε, ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν, προ, δεν πρόκειται να τα ακολουθήσουν. Και το σέβομαι αυτό και έχω και ιδιαίτερο θαυμασμό για τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους που ε, ύψωσαν τη φωνή τους εναντίον αυτών των γεγονότων. Και ελπίζω ότι θα ενδυναμωθεί η δημοκρατία στη ΣΥΠΑ συνάγοντας τα αναγκαία συμπεράσματα από τα όσα συνέβησαν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κυρία Χολμάιερ. Για τρία λεπτά εξ ονόματος Σοσιαλιστικής Ομάδας, ε, Τάνια Φαγιόν παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω ότι η συζήτηση που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή πράγματι θα πιάσει τόπο και ζητώ συγγνώμη που θα μιλήσω με κάθε ειλικρινία αλλά το θεωρώ απαραίτητο. Της ένας κρατούμενος τοποθετήθηκε σε ένα πολύ μικρό κλουβί το οποίο κρεμάστηκε τελικά και ο κρατούμενος παρέμεινε εκεί κρεμασμένος στο σιδερένιο κλουβί λόγω του ήλιου ή του κρύου και μετά είχαμε άλλους κρατούμενους που κρεμάστηκαν και είχαμε ε, διά του ορθού μέσω αντικειμένων, εχμηρών και ούτω καθεξής. Βλέπετε περιστατικά. Ε, αυτά τα πράγματα τα μάθαμε στο σχολείο για άλλες περιπτώσεις που αποτελούν μέρος της ιστορίας. Σε βασανιστήρι ένας κρατούμενος πέθανε από υποθερμία γιατί είχε αλυσοδευτεί σε γυμνός σε τσιμεντένιο πάτωμα. Παρακαλείστε να, μιλήστε να μιλάτε πιο αργά, λέει ο πρόεδρος. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ, απαντάει ο μελίτρια. Όλα αυτά μας υπενθυμίζουν τεχνικές μεσαίωνα, όμως δεν συνέβησαν το μεσαίωνα. Είναι η μέθοδοι ενισχυμένης ανάκρισης, τις οποίες προσέφηκε η CIA και έγιναν τον 20ο αιώνα. Και μάλιστα μια διαφορά εξίσου σημαντική είναι η εξής το 20ο αιώνα και το 19ο αιώνα ένα σωρό συμβάσεις ε, υπογράφησαν ε, συμβάσεις για τα δικαιώματα του παιδιού, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ούτω καθεξής και κυρώθηκαν σε όλο τον κόσμο. Οι ΙΠΑ έχουν υπογράψει σύμβαση κατά των βασανιστήριων και απαγορεύονται τα βασανιστήρια ακόμα και σε έκτακτες περιπτώσεις. Ζητώ συγγνώμη που σας ανέφερα τόσο φρικαλές λεπτομέρειες και που χρησιμοποιώ τον όρο «εμείς» γιατί το κάνω όμως διότι και εμείς είμαστε, πρέπει να κατηγορηθούμε για όλα αυτά. Εφτά χρόνια έχουμε περάσει από τότε που έχουμε μάθει ε, για τέτοιου είδους πτήσεις και για τέτοιου είδους πράγματα και οι ευρωπαϊκές χώρες συνεχίζουν να κρύβουν την αλήθεια. Δεν υπήρξε λογοδοσία, ούτε αποδόθηκαν ευθύνε. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ο αγώνας εναντίον της τρομοκρατίας δεν αποκλείει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε το αντίστροφο και τα θύματα πολέμου δικαιούνται δικαιοσύνη. Τα βασανιστήρια είναι ανήθικα και απαράδεκτα η συμμετοχή της Ευρώπης σε οποιαδήποτε μορφή παράνομες δραστηριότητες ε, της CIA είναι κάτι το επονίδιστο. Δεν αξίζουμε τη λέξη δημοκρατία. Δεν αξίζουμε τις αξίες που υποτίθεται ότι επικαλούμαστε. Απαιτούμε να γίνει πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και να υπάρξουν σαφείς απαντήσεις από πλευράς κρατών μελών. Η ασυλία, η ατιμορρησία είναι απαράδεκτη. Να υποκρινόμαστε ότι τίποτα δεν συνέβη και ότι δεν είναι δικό μας θέμα, δεν εμπλακόμαστε, αυτό είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να έχουμε αποτελεσματική δημοκρατία δημοκρατική εποπτεία στο έργο των υπηρεσιών πληροφοριών στις κατατόπους χώρας. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα ξαναγίνουν τέτοια πράγματα στην Ευρώπη ποτέ ξανά. Αγαπητοί συνάδελφοι, ορισμένε φορέ είναι πολύ δύσκολο να δεχθεί κανεί την αλήθεια, αλλά αξίζουμε να μάθουμε την αλήθεια και έχουμε την υποχρέωση να την ε, διαδώσουμε για να τη μάθουν και οι πολίτε μα. Πρέπει να κοιτάξουμε την αλήθεια ματά για να αποφύγουμε να είμαστε εμείς τους οποίους θα γίνουν τα βασανιστήρια αύριο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για την επόμενη ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών για δύο λεπτά μας μάκερ. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι όπως όλοι γνωρίζετε. Η Ευρωβουλή πάντα με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούσε τα θέματα των συλλήψεων και των φυλακίσεων από την CIA καθώς επίσης και της μεταφοράς των παράνομα κρατούμενων αυτών στην Ευρώπη από τη CIA. Έξι ψηφίσματα συνολικά εγκρίθηκαν από το Ευρωκοινοβούλιο κατά το παρελθόν για αυτό το θέμα. Τώρα, σε σχέση με την Αμερικανική Γερουσία και την έκθεση αυτή, που αφορά και ευρωπαϊκά κράτη που αναφέρθηκαν, όπως για παράδειγμα την Πολωνία, όπου υπήρχαν τέτοιες φυλακές ε, κράτησης ε, των παράνομα κρατούμενων ε, και όπου βοηθήθηκε η CIA. Το συμπέρασμα αυτής της έκθεσης ποιο είναι, Πρέπει να αναγνωρίσουμε εμείς οι ίδιοι το τι έκανα, κάναμε εμείς οι Ευρωπαίοι σε σχέση με τις αρχές και αξίες ε, της ε, ίδιας της Ευρώπης. Όμως ε, πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι αρχές και αξίες και να είναι σεβαστές από εμάς τους ίδιους και από τους συμμάχους μας. Δεν είναι δυνατόν να αναφέρονται μόνο ως αξίες, αλλά πρέπει να είναι σεβαστές. Είναι απόλυτα αναγκαίο να υπάρξει μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ της ελευθερίας και της ασφάλειας. Και πρέπει να πούμε ότι οι εξτρεμιστές στη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν κατάφεραν να ενισχυθούν και να ασκήσουν την επιρροή τους Τώρα, σε σχέση ε, με την υπονόμευση της ίδιας ε, της αξιοπιστίας και του κύρου της Ευρώπης, είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα. Πρέπει να είναι σεβαστές οι αρχές και τα δικαιώματα. Και σε μια πολιτική κατά της τρομοκρατίας από πλευράς Ευρώπης πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα του ανθρώπου και να διασφαλίζεται και η εμπιστοσύνη των πολιτών μας ε, στο δημοκρατικό μας σύστημα η ε, Ευρώπη με την υποστήριξη ε, του προγράμματος της CIA υπονόμευσε αυτή την αξιοπιστία των πολιτών της ε, και δεν είναι δυνατόν να παίζουμε τον δικαστή όταν εμείς οι ίδιοι είμαστε ένοχοι. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια για δυόμιση λεπτά, Σοφίν Φέλτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω την ε, γερουσιαστή Φέινστάιν για την επιμονή της και για το ότι πρόθεσε αυτή την έκθεση στην ε, Γερουσία. Η κυρία Χολμάγερ είπε πολύ σωστά ότι μας, όλα αυτά μας θυμίζει ότι η διαφορά μεταξύ δημοκρατίας και δικτατορίας είναι η λογοδοσία και το ηθικό κύρος. Και κανένας μας δεν είναι ε, στο απειρόβλητο Όλοι έχουμε τέτοιε τάσει ε, γενό. Αυτό που μα κάνει να διαφέρουμε είναι ότι λογοδοτούμε και ότι δεν υπάρχει ατιμορρησία σε μια δημοκρατία. Ε, με μεγάλη χαρά λοιπόν ακούω όλου του συναδέλφου από όλε τι πολιτικέ ομάδε που τονίζουν ότι πρέπει να υπάρξει λογοδοσία και ότι η Ευρώπη πρέπει η ίδια να αναγνωρίσει το ρόλο που έπαιξε σε αυτό το πρόγραμμα τη CIA. Γιατί μπορούμε να στελιτεύουμε του Αμερικανού, ε, αλλά και η Ευρώπη υποστήριξε το πρόγραμμα τρομοκρατία τη ΕΠΑ. Σε όλε τι πλευρέ του. Και χαίρομαι που επιτέλου το παραδέχτηκε η Πολωνία. Αλλά το παραδεχτούν και οι υπόλοιπε χώρε. Γιατί μην το ξεχνάμε, πολλά κράτη-μέλη είναι ε, στενοί σύμμαχοι ε, των ε, Ηνωμένων Πολιτειών. Και το Κοινοβούλιο εξέφρασε την υποστήριξή του πολλές φορές. Με εντύπωση ακούω ε, καταρχάς τις κοινοτοπίες της Ιταλικής Προεδρίας. Η Ιταλία είναι η χώρα η οποία δίωξε πράκτορες της CIA. Τους διώξατε και τους καταδικάσατε. Η Ιταλική Προεδρία θα επιμείνει σε, σε εκδόσεις, ούτως ώστε να εκδοθούν αυτοί οι άνθρωποι και να δικαστούν. Κύριε, κύριε Ομπάμα, όχι, δεν θα σταματήσουμε μέχρι οι υπεύθυνοι να συρθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Γι' αυτό είμαστε δημοκράτες, εμείς και άλλοι δεν είναι. Και μία ερώτηση που έχω εδώ είναι, διάβασα μία δήλωση στον τύπο από τον επικεφαλής του Κέντρου Πληροφοριών, που είναι ένα ειδο ε, σκοτεινού εμβριο, ε, έτσι, μυστικής υπηρεσίας ας πούμε. Και είπε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν λάβαμε πληροφορίες μέσω των βασανιστήριων. Παρακαλώ, Δηλαδή, ένας φορέας Ευρωπαϊκής Ένωση πληρώνεται με ευρωπαϊκό χρήμα, επεξεργάζεται πληροφορίε που μπορεί να έχει πάρει από τρίτε χώρε που μπορεί να έχει πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε πάρει από βασανιστήρια. Πρέπει να μάθουμε, πρέπει να πάρουμε απαντήσεις για τη φύση και τις δραστηριότητε. Ερωτήσεις που έχουμε υποβάλει κατά επανάληψη και εμείς θα πρέπει να ε, ασκούμε το δικό μας έλεγχο σε αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Δεχόσαστε ε, μία μπλε κάρτα τον κύριο Καρίμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι, κυρία Σόφη, ε, κυρία Σόφη Μπέλ, που δεχτήκατε την ερώτηση. Συμφωνείτε μαζί μου ότι αυτά που ακούσαμε από το Συμβούλιο σήμερα, ενώ ακούγονται πολύ γλυκά, στην πραγματικότητα είναι πολύ λίγα και ακούγονται πολύ αργά. Το 2005, εγώ ήμουν εδώ σε αυτή την αίθουσα και ήταν η Προεδρία του Συμβουλίου, τη είπα δε εκείνη τη μέρα ότι τα παράνομα κέντρα κρατήσεων υπήρχαν στην Ευρώπη. Δεν μα απάντησαν τίποτα τότε. Δεν μα είπαν ότι θα ερευνήσουν το θέμα. Και ο υπουργό τη Βρετανική κυβέρνηση που ήταν παρόν εκείνη τη μέρα στη θέση του Προεδρεύοντο, με αγνώρισε εντελώ. Συμφωνείτε λοιπόν ότι περαιτέρω έρευνε θα πρέπει να διενεργηθούν για να δούμε αν είναι σωστό οποιοδήποτε, το οποιοδήποτε υπουργό ε, ξέρει κάτι να κρύβεται πίσω από, την, πίσω από την, τον τίτλο ας πούμε, της Προεδρίας του Συμβουλίου και να μην δίνει πληροφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, λέει η κυρία Ιντβέλτ, συμφωνώ μαζί σας. Δεν αρκεί το Συμβούλιο, ούτε οι Ιταλοί Υπουργοί βεβαίω, ή οι κυβερνήσει των κρατών μελών να κάνουν δηλώσει για το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαίωμα, τι ε, διεθνεί συμβάσει και που έχουμε κτλ. Και τότε είχαμε νόμου. Αλλά δεν έγινε σεβαστή, παρακαλώ και δεν αρκεί. Δεν είναι καλό αυτό που μας λέτε, καλό και αρκετό. Αυτοί που παραβιάζουν τις, ε, τους κανόνες, ακόμα και να κυβερνήσει, θα πρέπει να διώκονται. Επομένως, ναι κύριε Καρύμ, συμφωνώ μαζί σας. Ευχαριστώ. Για την αριστερά, για 1,5 λεπτό τώρα, η κυρία Κολύρια Ευχαριστώ. Εκατοντάδες σελίδες φρίκης ε, τιμωρίες βασανιστήρια και σε ε, τμήματα του σώματος ε, σεξουαλική βία βλέπουμε ότι ατέλειωτες ώρες ε, δεν τους άφηναν να κοιμηθούν τους ε, βούταγαν στο νερό waterboarding όλα αυτά είναι τα στοιχεία της χειρότερης δικτατορίας που δίκαια καταδικάζουμε και σε διαφορά με, αυτις, με αυτές με αυτές δικτατορίες δημοσιεύουν οι τα στοιχεία αυτής της έκθεσης. Όμως έχουμε και την ε, σύμβαση καταδίκης και απαγόρευσης ε, των δικαστηρίων και βλέπουμε εδώ ότι συστηματικά δικασ... Ε, βασανιστήρια επιτρεπόντουσαν. Αυτό δείχνει τη βαθιά ηθική κρίση στις είπα που επιτρέπει να γίνονται τέτοια πράγματα. Δεν λειτουργούν τα βασανιστήρια κυρίες και κύριοι πουθενά. Όποιος η βασανιστήρια δεν μπορεί να διακριβώσει, να βοηθήσει να διακριβωθεί τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Και ε, δεν επαρκεί εδώ η κριτική και η καταδίκη. Πρέπει να απαγορευτούν τα βασανιστήρια παντού. Πρέπει νομικά να τα επεξεργαστούμε όλα αυτά. Και χαίρομαι ότι ο Γκρέγκορ Γκίζη στην Ομοσπονδιακή Γερμανική Βουλή ε, κατέθεσε ε, καταγγελία και κατηγορία εις βάρος του George Bush. Πρέπει να αποσαφινιστούν τα τι έγινε, όσα έγιναν με την εμπλοκή ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών από τα ευρωπαϊκά κράτη σε συνεργασία με την CIA. Πρέπει να πάψουν να υπάρχουν μυστικές κρυφές φυλακές και πρέπει να μην έχουν δικαίωμα να ασκούν αυτή την εξουσία. Ευχαριστώ. Για δυόμιση λεπτά στη συνέχεια θα λάβει τον λόγο για τους πρασινούς η Εύα Ζολή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, Κατά την ακρόασή σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προς μεγάλη μου έκπληξη, δηλώσατε ότι δεν γνωρίζατε την υπόθεση τότε. Διαπιστώνω με μεγάλη χαρά τώρα ότι σήμερα τη γνωρίζετε. Ωστόσο, ας το αναγνωρίσουμε. Δεν υπάρχει τίποτα το καινούριο που μαθαίνουμε στην έκθεση της Αμερικανικής Γερουσίας που εκτείνεται σε 600 σελίδες. Έχουμε επιβεβαίωση, επιβεβαίωση της συνεργασίας των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και το ότι υπήρχαν φυλακές και κέντρα κράτησης της CIA σε ευρωπαϊκό έδαφος. Επιβεβαιώνει η έκθεση ε, της Γερουσίας στην προσφυγή στα βασανιστήρια. Επιβεβαιώνει το ότι οι δράσεις των υπηρεσιών ε, πληροφοριών θα πρέπει να πλαισιώνονται αυστηρά να εποπτεύονται και ε, να τιμωρούνται οι μη ε, ένομες, σύνομες πράξεις. Και δεν θα πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα να θυσιάζονται στο όνομα του απαραίτητου αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Η δημοσίευση αυτής της έκθεσης μας καλεί να κινητοποιηθούμε έτσι ώστε να οικοδομήσουμε πραγματικά ε, δικαιοσύνη σε διεθνές επίπεδο. Το εύρος των εγκλημάτων μας υποχρεώνει να υιοθετήσουμε τόλμη στο νομικό επίπεδο. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καλείται να αναλάβει δράση. Ορισμένοι ηθήνοντες Ευρωπαίοι έχουν συνεργαστεί άμεσα σε αυτό το πρόγραμμα και γι' αυτό θα πρέπει να αναλάβουν δράση για τη διαφάνεια και ε, τα γεγονότα υπάρχουν, μιλούν από μόνο τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να διευκολύνουν την άσκηση δικαστικών διώξεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλει να συνεχίσει το διερευνητικό του έργο υπέρ της διαφάνειας έτσι ώστε να λάμψει η αλήθεια. Πρέπει να οργανώσουμε ακροάσεις, πρέπει αντιπροσωπείες της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών να μεταβούν σε αυτά τα κέντρα ε, κράτησης, τα κρυφά και τα μυστικά τα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταστρατηγήθηκαν. Τα άρθρα 4 και 6 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν κατά τη γνώμη σας, δεν θα πρέπει να εφαρμοστούν οι απαραίτητες κυρώσεις. Τέλος, να υπενθυμίσω ότι οι τρομοκράτες το μόνο που επιθυμούν είναι η κατάρρευση του αξιακού συστήματος το οποίο πρεσβεύει η δημοκρατία. Ε, Υιοθετώντας μεθόδους τις, τους, τις οποίες απαγορεύει ο νόμος, συνεπικουρούμε τους τρομοκράτες. Θα πρέπει να έχουμε διαφάνεια, ε, να αποκαλύψουμε την αλήθεια και να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Και αυτό δεν θα διευκολύνει τους τρομοκράτες, κάτι το οποίο κακώς φοβούνται κάποιοι. Αντιθέτως θα ενισχύσει τις αξίες μας ε, και θα υπάρχει ενισχυμένη δημοκρατία και όχι ενισχυμένη ανάκριση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. <clears throat> για την Ευρώπη της Άμεσης Δημοκρατίας για 1,5 λεπτό. Λάουρα Φεράρα παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο πτυχές που συνδέονται με την έκθεση της Αμερικανικής Γερουσίας για την προσφυγή στην, στο βασανιστήριο, στα βασανιστήρια από τη CIA. Καταρχάς πρέπει να σκεφτούμε. Πρέπει να σκεφτούμε την δυνατότητα άσκησης αυτοκριτικής των δημοκρατικών αμερικανικών ε, θεσμών. Ε, και από την άλλη το θέμα της ε, εθνικής ε, ασφάλειας. Βλέπουμε αυτό το πνεύμα των Αμερικανικών αρχών. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας εμποδίσει να καταδικάσουμε οποιαδήποτε μορφή βίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άσκησης βίας και αγνόησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων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 Ενάμιση λεπτό είχατε από την ομάδα σας. Εντάξει, φτάνει. Ολοκληρώσατε. Από τους μη εγγεγραμμένους, η συνάδελφος Κριστίνα Μορβάη. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερος διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά εκφράζει την κατάπληξή του με την καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς πλευρά Επιτέλους, ή τα βασανιστήρια ή η κράτηση η δίκη είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί. Ωστόσο, πριν από λίγους μήνες είχαμε την υπόθεση Snowden και ε, το σκάνδαλο με τις μυστικές έρευνες κτλ. Αυτά ε, μας απασχόλησαν και στη συνέχεια σε διάφορους πολέμους άμαχοι βρήκαν το θάνατο πάλι με δράση Ηνωμένων Πολιτειών. αναρωτιέμαι όμως και απορώ αν τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι τόσο πια θυμωμένο με τις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί θέλουμε τόσο πολύ την Αμερικανική φιλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δουλεύει στενά, συνεργάζεται με τη ΣΥΠΑ και σε οικονομικό επίπεδο και στα υπόλοιπα επίπεδα. Προσπαθούμε να πετύχουμε μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με τη ΣΥΠΑ η οποία γίνεται αντικείμενο διαπραγματεύση και κλεισμένων των θυρών, η Ευρωπαϊκή Ένωση από εκεί και πέρα ανταποκρίνεται και αντιδρά στι ε, ε, εγκλήσεις και στα αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και τελικά υπάρχει ένας, ένα ψυχροπολικό μικρό κλίμα που έχει εγκαθιδρυθεί με τη Ρωσία και υπάρχει και φόβος ότι αυτό θα μεταφραστεί ε, και θα επεκταθεί ε, σε πλήρης καταστάσεις σύγκρουσης με τη Ρωσία. Δεν θα πρέπει όλα αυτά να μας απασχολήσουν. Ε, εμείς στην Ουγγαρία έχουμε μεγάλη εμπειρία από το ψυχρό πόλεμο και φοβόμαστε την προοπτική ενός αληθινού πολέμου. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε κυρία Μορβάη. Τώρα οι επιμέρου ευρωβουλευτέ. Θα είμαι πιο αυστηρός τώρα με το χρόνο. Έχουμε μακρύ κατάλογο αγοριτών. Ο πρώτο, Κρίστιαν Πρέντα. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η χρήση των βασανιστήριων από τη CIA είναι ένα θέμα που πόλωσε την κοινή γνώμη στι ΗΠΑ εδώ και χρόνια. Η δημοσίευση της έκθεσης της ε, Γερουσίας την περασμένη εβδομάδα επιβεβαίωσε το χάσμα που υπάρχει, την πόλωση που υπάρχει και στην αμερικανική πολιτική τάξη. Οι δημοκράτες και οι ρεπουμπλικάνοι είναι βαθιά διαιρεμένοι σε ό,τι αφορά διάφορα θέματα. Φερρυπίν, η έκθεση αντικατοπτρίζει σωστά και πιστά αυτά που συνέβησαν. Δεύτερον, η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε ήταν σωστή αυτή η έκθεση έπρεπε να δημοσιευτεί δεδομένων των πιθανών επιπτώσεων στην ασφάλεια. Όλα αυτά τα προβλήματα έχουν ακουστεί, έχουν αναφερθεί και ακόμα δεν έχει δοθεί σαφής απάντηση στις ΗΠΑ. Δεν υπάρχει μία και μόνη απάντηση που μας έρχεται από τις ΗΠΑ. Θα ήθελα να τονίσω ότι εγώ προσωπικά συμφωνώ αρκετά μετά όσα είπε ο Τζον Μακκέιν, ο ρεπουμπλικάνος ε, γερουσιαστής που ζήτησε να δημοσιευθεί η έκθεση και που επέκρινε τη CIA και που η δήλωσή του νομίζω ήταν πάρα πολύ συνετή. Είπε, πήγαμε, κάναμε λάθη, δεν, κάναμε, δεν κινηθήκαμε σωστά, θα πρέπει να διορθώσουμε τα, άλλη και δεν θα ε, τα λάθη και δεν θα πρέπει να τα επαναλάβουμε. Σήμερα κανένας δεν μπορεί να πει ότι οι πρακτικές αυτές, οι οποίες τον αναφέρονται στα, στην έκθεση αυτή, συνεχίζονται. Είναι κάτι το οποίο σταμάτησε. Σταμάτησαν αυτές οι ανακρίσεις από τον Ομπάμα το 2009. Και υπάρχει μια σαφής θέληση στις ΗΠΑ να διερευνηθούν όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι είναι αυτό το βασικό πράγμα που πρέπει να κρατήσουμε. Όταν μια πολιτική οντότητα αναλύει τα δικά της λάθη, αυτό είναι πάρα πολύ υγιές. Για τρία λεπτά η συνάδελφος είπε, παρακαλώ. Όποιος ακούει τα λόγια του Συμβουλίου μπορεί να αποκομίσει την εντύπωση ότι σε εμά όλα πάνε καλά λέει. Μεγάλο σφάλμα αυτό. Τα βασανιστήρια της CIA είναι φρικτά εγκλήματα όπως στα οποία συμμετείχαν και ήταν συνένοχα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συστηματικά και παραβιάζοντας κάθε διεθνή αρχή και αξία συστηματικά βασανιζόντουσαν άνθρωποι από την CIA και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυριζόταν η CIA ότι αξιόλογα στοιχεία έπαιρνε από τα βασανιστήρια για την αποτροπή τρομοκρατικών πράξεων. Ψέμα αυτό. Αλλά ανεξάρτητα από όλα αυτά, τα βασανιστήρια δεν μπορεί να είναι μέσο στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Είναι τα βασανιστήρια τα ίδια έγκλημα και παραβιάζουν την, τον πυρήνα των αρχών και των αξιών μας. Αυτό μας διαφοροποιεί από τους φονταμενταλιστές και τους εξτρεμιστές και πρέπει στην πρόληψη να δράσουμε και στην καταπολέμηση τρομοκρατικών πράξεων να μιλήσουμε με άλλη γλώσσα και να μην χρησιμοποιούμε τη γλώσσα της βίας. Διαφορετικά δίνουμε επιχειρήματα στους εξτρεμιστές να απορρίπτουν και να μισούν τα δημοκρατικά καθεστώτα μας, τη δημοκρατία. Δεν είναι μόνο θέμα ηθικής αυτό. Είναι απλά θέμα διεθνούς δικαίου. Τα βασανιστήρια δεν επιτρέπονται ποτέ πρέπει πάντα τα βασανιστήρια, πάντα από όλα τα κράτη να καταδικάζονται και να διώκονται. Είναι έσχος, ντροπή για την Ευρώπη ότι ευρωπαϊκά κράτη έκλεισαν και τα δυο τους μάτια όταν υπήρχαν οι παράνομες μεταφορές κρατουμένων και υπήρχαν φυλακές παράνομες στην ίδια την Ευρώπη. Ήδη το 2007 το Ευρωκοινοβούλιο απέτησε ε, ε, ευρύτερες διακριβωτικές ε, έρευνες χωρίς αποτέλεσμα όμως. Εκείνοι οι οποίοι πολίτες, πολίτες που ήταν ακόμα και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συλλαμβάνονται χωρίς καταδικαστική απόφαση δικαστηρίων, να κρατούνται σε παράνομες φυλακές και να βασανίζονται. Την προηγούμενη εβδομάδα κιόλα ανώτεροι αξιωματούχοι της Πολωνίας ε, ε, επιβεβαίωσαν την ύπαρξη αυτών των μυστικών φυλακών. Οι εθνικές κυβερνήσεις μόνες τους προφανώς δεν είναι σε θέση να κάνουν κάτι γιατί έχουν εμπλακεί, ενεπλάκησαν σε αυτά τα εγκλήματα οι ίδιες. Χρειάζονται μηχανισμοί από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε τέτοιου είδους πράξεις να μην παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Δείχνουν όλα αυτά το τι συμβαίνει όταν παρακάμπτεται ένα κράτος δικαίου και δημιουργείται μια, ένα καθεστώς τρομοκρατίας. Κανείς δεν προστατεύεται η ίδια η δημοκρατία μας συνολικά απειλείται και υπονομεύεται. Αδιαφορούν όλοι οι υπεύθυνοι αν εμείς ως Ευρωπαίοι θα, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Εμείς όμως πρέπει να κάνουμε κάτι και πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας συνδράμει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε και ευχαριστώ που τηρήσατε ακριβώς τον χρόνο που είχατε. Για ένα λεπτό τώρα ο κύριος Κρασνογεύσκη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε το γεγονός ότι στην πολωνική επικράτεια ε, είναι πιθανό να έχουν διαπραχθεί αυτά τα βασανιστήρια ε, είναι κάτι που καταδίκασε απερίφραστα η πολωνική κοινή γνώμη. Παρόλο που κάποιοι προσπάθησαν να δικαιολογήσουν αυτές τις πρακτικές και παρόλο που ήταν ύποπτοι οι κρατούμενοι για τη δολοφονία χιλιάδων ανθρώπων. Σήμερα θα δημοσιευθεί μια ανοιχτή επιστολή με την υπογραφή πολύ σημαντικών προσωπικότητων της Παλωνίας καταδικάζοντας αυτές τις πρακτικές. Θέλω να σας εφιστήσω την προσοχή όμως στο θέμα των διπλών προτύπων, των διαφορετικών μέτρων και σταθμών και στο θέμα της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ συμμάχων. Εάν η CIA δεν είχε διενεργήσει τέτοια ανάκριση ε, στην επικράτεια των ΗΠΑ γιατί σεβάστηκε τον νόμο ε, των ΗΠΑ, ωστόσο δεν σεβάστηκε την αντίστοιχη πολωνική νομοθεσία. Και δυστυχώς οι θύνοντε οι Πολωνοί δεν σεβάστηκαν το γεγονός ότι η Πολωνία είναι κυρίαρχο κράτος. Δυστυχώ, ε, καταχράστηκαν τις εμπιστοσύνη μας και γι' αυτό η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό, Σεσίλια Βίξτρομ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πραγματικά μας ανησυχεί και με φρίκη βλέπουμε το τι συνέβη από τα στοιχεία της έκθεσης της Γερουσίας για τα βασανιστήρια της CIA που ήταν φρικαλαιότητες. Ποιες έννοιες πρέπει να χρησιμοποιηθούν. Φρίκη για τον τρόπο με τον οποίο θέλησαν κιόλας να διαψεύσουν αυτά τα στοιχεία υπεύθυνοι της CIA κατά το παρελθόν. Ατιμορρησία έναντι αυτών των τρομερών της τρομερής παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Και όλα αυτά εξ ονόματος των είπα για την ασφάλεια λέει. Και όπως αναφέρθηκε, όταν δει κανείς ε, τα, τις συνέπειες, ε, τις επιπτώσεις ε, των βασανιστήριων βλέπει κανείς ε, ότι δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Άσχετα από αυτό πρέπει να επαναλάβουμε και να πούμε τα βασανιστήρια δεν επιτρέπεται να διεξάγονται υπό καμία πρόφαση και πρόσχημα. Διεθνώς απαγορεύονται και υπάρχει και σύμβαση που τα απαγορεύει και πρέπει να ισχύει για όλους αυτό. Από την έκθεση βλέπει κανείς ότι κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Σουηδία, η Μεγάλη Βρετανία, η Ρουμανία συνεργάστηκαν κιόλα με τις με τη CIA. Και οι ίδιες οι αρχές ε, ασφάλειας ε, των ΗΠΑ συνέλαβαν και ε, φυλάξαν ανθρώπους χωρίς δικαστικές, καταδικαστικές δικαστικές αποφάσεις και, και από την ίδια τη Σουηδία υπό απαράδεκτους όρους και συνθήκες. Τώρα δεν μπορούν να, να διαψευστούν αυτά περαιτέρω. Πρέπει να ακουστεί η αλήθεια και πρέπει να πούμε την αλήθεια. Αυτό θα μας απελευθερώσει από την ενοχή, την ενοχή μας και πρέπει εκείνοι που είναι υπεύθυνοι να προσαχθούν στη δικαιοσύνη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Άντερσον παρακαλώ. I know you agree with me that... Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι τα βασανιστήρια είναι ανήθικα, παράνομα και πρέπει πάντα να καταδικάζονται. Και εξάλλου και με τις ε, στρατιωτικές ε, δυνατότητες ε, ανακρίσεων αναφέρομαι σε σχέση με τα όσα είπε ο Τιμ Κόλλιν στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που υπηρετούσα οι κανόνες ανάκρισης μετατράπηκαν από πλευράς των νομικών πλαισίων. Φτάσαμε στο σημείο όπου χάσαμε την αποτελεσματικότητά μας μέσα στο πλαίσιο αυτών των ανακρίσεων. Έχετε λίγο χρόνο και αν βιάζεστε τόσο πολύ δεν είναι δυνατόν οι διερμηνείς να σας παρακολουθήσουν ε, υπενθυμίζει ο πρόεδρος. Παρακαλώ το λάβετε υπόψη αυτό. Είναι η τρίτη φορά σήμερα. Αυτά τα οποία αναφέρετε θα πρέπει να είναι κατανοητά στους άλλους. Μπορείτε να επιβραδύνετε. Καταλάβατε την ερώτηση. Όχι. Ε, ε λοιπόν προχωρούμε στη συνέχεια. Θα έχετε μια ευκαιρία να απαντήσετε. Με ιδιαίτερη χαρά να απαντήσω η κτηνοδία, η ομότητα των μεθόδων σε σχέση με τα όσα έγιναν είναι απαράδεκτη και τα κράτη, τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να συνέρθουν ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Τι έγινα στη δική σας χώρα, τι συνέβη στη δική μου χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να αποκαλυφθεί. Να την πούμε τώρα. Πρέπει να πάψει πια, να τερματιστεί η ατιμορρησία, ακόμα και στην Ευρώπη την ίδια. Ευχαριστώ. Thank you very Σας ευχαριστούμε πολύ. Για 1,5 λεπτό στη συνέχεια, Ματίνα Άντερσον, παρακαλώ. Η πρόσφατη έκθεση της Γερουσίας για τις τεχνικές της CIA δείχνει ε, ποιες είναι τεχνικές των Αμερικανών, ε, βασανιστήρια κτλ. Οι πέντε τεχνικές που χρησιμοποίησε η Βρετανική κυβέρνηση για να βασανίσει 14 Ιρλανδούς ε, επί χρόνια ήταν ίδιες. Η Ιρλανδική κυβέρνηση έσυρε τη Βρετανική κυβέρνηση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ήταν η πρώτη φορά που ένα κράτο μέλο έσυρε ένα άλλο κράτο μέλο σε δικαστήριο. Έγινε το, το 1978 αυτό. Όμω το δικαστήριο είπε ότι πέντε ε, τακτικέ ήταν ε, απάνθρωπη μεταχείριση αλλά όχι βασανιστήριο. Και αυτές οι τεχνικές στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στο Γουατάναμο Μπέι ε, τις, υποστήριξαν οι Αμερικανοί, χρησιμοποιώντας κουκουλοφόρους άντρες. Οι 14 κουκουλοφόροι στην πραγματικότητα ήταν δήμοι. Αυτές οι τεχνικές όμως χρησιμοποιήθηκαν και στο Βρετανικό, ε, από την Βρετανική κυβέρνηση και τις επικύρωσε τα υψηλότερα κλιμάκια της Βρετανικής κυβέρνησης. Θα πρέπει το δικαστήριο να αναθεωρήσει την άποψή του γιατί ε, θα πρέπει ε, να καταδικαστεί η Βρετανική κυβέρνηση και να απολογηθεί για τις τεχνικές αυτές. Και νομίζω το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για την Αμερική. Συνάδελφοι, έχουμε ένα θέμα στη μερίσια διάταξη. Θα πρέπει να μιλάτε εντός θέματος και όχι εκτός θέματος. Σαρτζεντίνη. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Τα βασανιστήρια τη CIA είναι το θέμα μας. Η έκθεση Feinstein μας αφυπνίζει πολύ βία στην Ευρώπη. Και αυτό είναι πολύ σωστό, γιατί στην ομάδα μου προσπαθήσαμε τους τελευταίους μήνες να βάλουμε στην ημερήσια διάταξη μία έκθεση που εμείς είχαμε ετοιμάσει και να ασχοληθούμε με τις εμπλεκόμενες ευρωπαϊκές χώρες που είχαν, που είχαν χρησιμοποιηθεί από τους Αμερικανούς. Γιατί χρησιμοποιήθηκαν ευρωπαϊκά εδάφη από τους Αμερικανούς. Όμως δεν υπήρχε πια ενδιαφέρον για κάτι τέτοιο. Όμως βλέπω ότι με τη σημερινή συζήτηση κάνουμε μια νέα αρχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, εμπλοκή των ευρωπαϊκών κρατών στα βασανιστήρια της ΣΥΑ. Ο κ. Παπαδάκης για ένα λεπτό είναι ο επόμενος ομιλητής. Τα βασανιστήρια της CIA δεν εκπλήσουν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι μυστικές υπηρεσίες τους μέχρι σήμερα έχουν πλούσιο ιστορικό από υπεριαλιστικέ επεμβάσεις, χούντες, πραξικοπήματα, άγρια βασανιστήρια, εμψυχρό δολοφονίε Αφροαμερικάνων. Η δε Ένωση πάει πολύ να αυτοπροβάλλεται ως ο τιμητής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. η κοινή εξωτερική πολιτική ασφάλειας και άμυνας η europol η Eurojustice, όλοι οι μηχανισμοί καταστολής της ευρωπαϊκής ένωσης και του νατο είναι εταίροι και σύμμαχοι της cia. τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης συνεργάζονται με τις ηνωμένες πολιτείες σε πολλούς τομείς καταστολής του εργατικού λαϊκού κινήματος επίσης στην κρατική και βιομηχανική κατασκοπία στις τηλεφωνικές και διαδικτυακές παρακολουθήσεις ενώ καλύπτουν τα απάνθρωπα βασανιστήρια. όλα αυτά δεν αποτελούν παραφωνία του καπιταλιστικού συστήματος αλλά το πραγματικό του πρόσωπο. στόχος τους είναι η υπεράσπιση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης ενάντια στον εχθρό λαό. αυτή είναι η δικτατορία των μονοπωλίων και οι λαοί μπορούν να πάρουν τις αποφάσεις τους για να την ανατρέψουν με τη δική τους εξουσία. έχουν τη δύναμη. Vielen Σας ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά ο συνάδελφος Σέλμαρ Μπρόκ τώρα, παρακαλώ. Ε, ε- κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε, βρίσκω ότι είναι μεγάλο επίτευγμα της Αμερικανικής Γερουσίας και ιδιαίτερα της Γερουσίας του Φάινστάιν η δημοσιοποίηση αυτής της έκθεσης. Αυτό τι δείχνει. Δείχνει σε αντίθεση με τα όσα συμβαίνουν στην Κίνα και στη Ρωσία ότι η ΗΠΑ είναι σε θέση τα λάθη που έκαναν οι, οι ίδιες οι ΗΠΑ να τα επανορθώσουν. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά κιόλα. μεταξύ μιας δικτατορίας και μιας δημοκρατίας. Δεν πρέπει κιόλας να υβρίζεται μια δημοκρατία γι' αυτό. Ωστόσο αληθεύει, αυτά τα οποία συνέβησαν είναι πραγματικά δικαιολόγητα και δεν υπήρχε κανένας λόγος, ε, δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να δικαιολογηθούν και είναι απόλυτα παράνομα. Είναι απάνθρωπα και πρέπει να κατακριθούν και να καταδικαστούν. Είναι απόλυτα σαφή όλα αυτά. Και εγώ ο ίδιος ε, είχα επισκεφθεί το Γουαντάναμο και τοποθετήθηκα σαφώς σε αυτό το θέμα, ότι είναι απαράδεκτα αυτά και ότι δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Σωστές αυτές οι επικρίσεις, αλλά όχι με υποκριτικό τρόπο να κατηγορούμε τη ΣΥΠΑ και να λέμε ότι είναι ο μεγαλύτερος ένοχος. Πρέπει να δούμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσχημα αλλά είναι συνέπεια τρομοκρατικών πράξεων που υπέστη ο Αμερικανικός λαός που υπέστησαν οι ΙΠΑ και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη και να το αναφέρουμε και το επαναλαμβάνω δεν μπορεί να υπάρξει απολογισμός ελευθερίας και ασφάλειας με τόσο λανθασμένο και στρεβλό τρόπο ώστε να μην είναι σεβαστά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Γι' αυτό ασκούνται επικρίσεις. Οι Αμερικανοί αποκαθιστούν τώρα τη σωστή αναλογία των πραγμάτων. Μπορούμε να ασκήσουμε επικρίσεις, αλλά πρέπει να κατανοήσουμε ακριβώς πώς και τι συνέβη. Και θέλω να πω και να εκφράσω με αυτό ότι είχαν το θάρρος οι Αμερικανοί με όλες τις συνέπειες να αναφέρουν το τι έγινε και να υπομισθούν τις ευθύνες. Αυτό διαφοροποιεί τη ΣΥΠΑ από πολλές δικτατορίες παγκόσμια και που θα πρέπει πραγματικά να λάβετε υπόψη το γεγονό γεγονός ότι φυλακίζονται από αυτές τις δικτατορίες άλλοι και εξακολουθούν να γίνονται όλα αυτά. Δέχεστε μια ερώτηση από συνάδελφο Ευρωβουλευτή, κύριε Μπρόκ. Mr. Page, you have the floor. Κύριε Φέιτ, έχετε τον λόγο παρακαλώ για την ερώτησή σας. Ma jagan härra Brocki τις απόψεις του κύριου Μπρόκ, έχω όμως μια ερώτηση που θα ήθελα να διατυπώσω Ποιους θεωρεί τους κινδύνους ο κύριος Μπρόκ στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Βλέπετε να υπάρχουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις ε, σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας από τα στοιχεία αυτής της ε, έκθεσης. Είδαμε τα φρικαλαία συμβάντα στο Πακιστάν πρόσφατα. Ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά. Κύριε Μπρόκ, ναι, για την έκφραση ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να αναγνωριστεί. Ωστόσο, η παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με την παραβίαση των δικαιωμάτων. Ασκούνται λοιπόν επικρίσεις, πρέπει να δούμε όμως τη σωστή συνάφεια των πραγμάτων. Ευχαριστώ. Κύριε Μπρόκ, ο λόγος σας έχει προκαλέσει και άλλες ερωτήσεις. Έχω άλλες δύο μπλε κάρτες από την κυρία Ίντφερτ και τον συνάδελφο Κάντης. Δέχεστε. Ε, τότε και οι δύο ερωτήσεις, η μία μετά την άλλη και η απάντησή σας ένα λεπτό στη συνέχεια. Παρακαλώ κυρία Ινφέλτ. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Χαίρομαι που ο συνάδελφος Μπροκ καταδικάζει την uh, χρήση των βασανιστήριων. Στο, στο παρελθόν είχε πει ότι ε, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι περιστάσεις κτλ. Είναι αλήθεια κύριε Μπροκ ότι παρότι μερικές φορές καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι περιστάσεις ε, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που δεν διώξαμε αυτούς τους ανθρώπους, ενώ θα έπρεπε να έχει υπάρξει λογοδοσία. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες μέχρι σήμερα. Και σε ό,τι αφορά τη δικαιοσύνη, οι Αμερικάνοι κλείδωσαν ανθρώπους στη φυλακή, όπως τον Τζον Κυριάκου, ε, που ήταν ε, υπάλληλος της CIA, στη φυλακή γιατί αποκάλυψαν διάφορα στοιχεία. Έκανε φυλακή ο άνθρωπο αυτό. Δεν είχαμε χρόνια ολόκληρα για να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε. Δεν συμφωνείτε με αυτό, παρακαλώ. Κύριε Μπροκ, σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σα. Εγώ ως φίλος τον είπα, δεν θα πρέπει να του ζητήσουμε να κλείσουν επιτέλους τον Καντάναμο Μπέι. Σα ευχαριστώ. Και άλλη μια ερώτηση. Η συνάδελφο Έρνστα αναφέρθηκε προσωπικά και παίρνει τώρα την μπλε κάτα για να θέσει την ερώτησή τη. Συμφωνώ οπωσδήποτε σε κάποια πράγματα μαζί σα κύριε Μπρόκ. Όμω ήθελα να θέσω την εξή ερώτηση. Δεν βρίσκεται ότι για αυτά Κάτι θα έπρεπε νομικά να γίνει. Νομικά μέτρα και πρωτοβουλίε θα έπρεπε να ληφθούν κατά εκείνων που παραβίασαν τα δικαιώματα του ανθρώπου με αυτέ τι πράξει και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Νομικέ δηλαδή συνέπειε. Πώ το βλέπετε. Σα ευχαριστώ. Έχετε ένα λεπτό κύριε Μπρόκ να απαντήσετε στι ερωτήσει. Μάλιστα. Ήταν σφάλμα κατά το παρελθόν αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί και να επανορθωθεί και πρέπει και να υπάρξει και δικαστική επανόρθωση σε σχέση με τις πράξεις αυτές. Όμως ε, δεν αλλάζει αυτό τα επιχειρήματα τα οποία εξέθεσα και θα πρέπει τώρα για την, τη διάλυση, το κλείσιμο του Γουαντάναμο πριν από 8 ή 10 χρόνια το είχα ζητήσει αυτό. Δεν πρέπει να το επαναλάβω. Πάντα το πίστευα ότι έπρεπε να κλείσει. Όμως πιστεύω ότι τα δύο μέτρα και σταθμά που έχουμε, ποια από τα κράτη μας ήταν πρόθυμα να δεχθούν κρατούμενους του Γκουαντάναμο όταν ζήτησαν οι Αμερικανοί να παραδοθούν σε ευρωπαϊκά κράτη αυτοί οι κρατούμενοι. Μόνο λίγες χώρες ήταν πρόθυμες κάποιους να δεχθούν από αυτούς τους κρατούμενους. Και έτσι έχουμε λοιπόν αυτή την επίφαση ηθικής που επικαλούνται κάποιοι υποκριτικά εδώ εις βάρος των Αμερικανών. Και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με αυτό το γεγονός. Δεν υπάρχει εδώ μια ε, προθεσμία παραγραφής αυτών των ε, εγκλημάτων σε σχέση με, τις, ε, με τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε στη συνέχεια για δύο λεπτά ο συνάδελφος Κλοντ Μωράη. Thank you, President. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα πράγμα θα πω ότι ο κύριο στο μόνο που έχει δίκιο είναι ότι και οι δύο συναντήσαμε την γερουσιαστή κυρία Φάινστάιν. Επέδειξε θάρρο τότε και πραγματικά επέδειξε μεγάλο θάρρος σε αυτό το θέμα. Η πέστη τεράστια πίεση κατάφερε να κάνει τα πάντα έτσι ώστε να προχωρήσει αυτή η έκθεση και ο κύριος Κοέλιο θα συμφωνήσει ότι ε, τώρα ε, επανέρχεται το θέμα ε, των εκθέσεών μας του 2006 για τις έρευνες και τις ανακρίσεις της CIA. Όλα αυτά τότε όμως ήταν τελείως διαφορετικά. Το 2006 όταν διερευνήσαμε τις δευτερογενείς πηγές και όχι τις πρωτογενείς πηγές που είχε στη διάθεσή της η Αμερικανική Γερουσία, εμείς λοιπόν όταν τα διερευνήσαμε όλα αυτά, όλες αυτές οι φρικαλές και βάρβαροι, βάρβαρες μέθοδοι βασανιστήριων κληθήκαμε να ασχοληθούμε με αυτά. Όμως οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές, ήταν πολύ έφραυστη και λεπτή η κατάσταση, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μας τότε και, ποια ήταν, και είχαμε και δυσκολίες στην έρευνά μας και καταλήξαμε στο εξή συμπέρασμα, το συμπέρασμα του Τζον Μακκέιν. Εάν καταλαβαίνετε τη διαφορά μεταξύ ανάκρισης και ε, φρικτών βασανιστήριων, καταλήξαμε στο ίδιο συμπέρασμα με τον Τζον Μακέιν, ότι δηλαδή ήταν εσφαλμένο αυτό, ήταν λάθος, ανήθικο και δεν έφερε νέα στοιχεία υπέρ του αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Όλοι αυτοί, ο Τζον Μακέιν και οι λοιποί, είναι ε, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν την ποιοτική διαφορά του να μην έχει καθόλου κανείς στοιχεία και πληροφορίες ή να έχει κακά, κακής ποιότητας στοιχεία και πληροφορίας. Ε, δεν έχουμε φτάσει στο τέλος. Αυτή τη στιγμή ε, φυτοζούν άνθρωποι στη βάση του Γουαντάναμο και ζητούν οι κυβερνήσεις τους να απελευθερωθούν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βασανιστεί, που ε, ε, κινδυνεύουν. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία. Έχει μόλις ξεκινήσει. Είναι δικοί μας πολίτες, πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διαβιούν σε φρικτές συνθήκες στο Γουαντάναμο και αλλού. Έχουν βασανιστεί. Τους θέλουμε πίσω να επιστρέψουν και θα πρέπει να τους εκπροσωπούμε. Ευχαριστώ. E, e, Έχετε μια μπλε κάρτα, κύριε Καν. Κύριε, από τον κύριο Καν. Κύριε το δέχεστε. Κύριε Καν, παρακαλώ. Τα μέλη που δεν ήταν εδώ το 2006 θα ήθελαν να μάθουν κάτι. Είπατε δύο πράγματα. Είπατε ότι δικαιωθήκαμε και ότι ήταν δύσκολο. Γιατί τα είπατε αυτά. Ευχαριστώ, γιατί ήταν δρακονικός. Να πω στους Ευρωβουλευτές και στον κύριο Κοέγιο, που ήταν πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής τότε, πολύ αποτελεσματικά. Ο Κλάουντιο Φάβα ήταν ο εισηγητής, Ιταλός, που είναι τώρα μέλος της Ιταλικής Βουλής. Ήταν βουλευτέ οι οποίοι ανέλαβαν πολύ δύσκολο καθήκον. Η αξιολόγησή μου είναι ότι οι τρεις μεγάλες έρευνες του Κοινοβουλίου, η έρευνα εσελών, η έρευνα για τις μασικές υποκλοπές και για τις μυστικές μεταφορές κρατουμένων πτήσεων, είπαν το ίδιο πράγμα, ότι έχουμε επαρκή κοινοβουλευτικό έλεγχο για τέτοιες ε, δράσεις. Ε, αυτός, η κοινοβουλευτική εποπτεία επιτρέπει να διερευνούμε τέτοιες πράξεις, τέτοιου είδους πράξεις που τώρα εξετάζουμε, που α, σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί βασανιστήρια κτλ. Γι' αυτό θα πρέπει τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου να πιστεύουν, να ενδιαφερθούν για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Πρόεδρος, έχουμε ακόμα μία μπλε κάρτα. Α, τον κύριο Κάριντον. Καρίμ. Το δέχεστε. Ευχαριστώ τον Κλωτ Μωράε για τη δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό επί χρόνια. Σας ρωτάω κύριε Μωράε, μία από τι μεγαλύτερε προκλήσεις που είχαμε είναι το να πάρουμε πληροφορίε από τι δικέ μα κυβερνήσει. Πιστεύετε ότι είσαστε ικανοποιημένο ότι είχαμε, μας αποκάλυψαν όλα τα στοιχεία από τις... Δηλαδή, οι κυβερνήσει των κρατών μελών μα τα αποκάλυψαν. Και αν όχι, πώ μπορούμε να ικανοποιηθούμε και να είμαστε σίγουροι ότι κανένα από του πολίτε μα θα αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση ποτέ πια. Φυσικά δεν υπάρχει πλήρη αποκάλυψη. Γι' αυτό η κυρία Φάινστάιν είναι πολύ γενναία. Εγώ και ο Μπρόκ την συναντήσαμε. Και μόλι τη συναντήσαμε, ε, συνειδητοποίησαμε πόσο γενναία είναι. Ε, αυτή η γερουσιαστή. Είμαστε βουλευτέ, ε, και ε, ασχολούμαστε με την έρευνα αυτή τη CIA. ξέρουμε πολύ καλά ότι και οι δικέ μα κυβερνήσει εμπλέκονται. Μερικέ φορέ ε, μέλη της κυβέρνησης α, προσπαθούσαν να μάθουν την αλήθεια. Φυσικά δεν υπάρχει πλήρης αποκάλυψη. Πρέπει να είμαστε ε, επίμονοι, γενναίοι και να μάθουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Μερικές φορές δεν μαθαίνουμε απευθείας αλλά από δεύτερο χέρι. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουμε. Χωρίς την λογοδοσία αυτή δεν φτάνουμε στην αλήθεια. Επίσης, υπάρχουν ακόμα Ευρωπαίοι πολίτες στη φυλακή. Ακόμα αθώοι απόλυτα ε, αθώοι και θα πρέπει να απελευθερωθούν. Γι' αυτό το θέμα αυτό είναι τόσο σωτική σημασία και όλοι οι βουλευτές ε, θα πρέπει να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους, αν μη τι άλλο. Ο κύριος ένα λεπτό. Ως επί πολλά χρόνια μέλος της Διεθνούς Αμνηστίας Amnesty International όπως και εσείς ε, έχω πραγματικά εκπλαγεί και με φρίκι διαπιστώνω το τι συνέβη από πλευρά των ΗΠΑ. Πρέπει όμως να υπενθυμίσω ότι οι ίδιοι Αμερικανοί ήταν εκείνοι οι οποίοι δημοσιοποίησαν αυτά τα πράγματα. Η Γερουσία ήταν αυτή που τα δημοσιοποίησε και και εκεί όπως και εδώ με κριτικό πνεύμα συζητώνται και αναλύονται αυτά τα οποία προκάλεσε και έκανε η Αμερικανική κυβέρνηση. Αυτό που με εκπλήσει είναι ότι εμείς πάλι έχουμε τους Αμερικανούς που κατηγορούμε. Θα ήθελα να υπάρξει μια συζήτηση για αυτά που έκανε η ρωσική μυστική υπηρεσία και έχει διαπράξει. Αυτό βλέπω να απουσιάζει εδώ. Και ως συνεισηγητής, συνεισηγητής της έκθεσης για την κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου πέρυσι πρόσεξα ότι σε αυτή την έκθεση πάντα ασχολούμαστε με πράγματα που είναι αξιοπερίεργο ότι στρέφονται τις περισσότερες φορές κατά των Αμερικανών. Καλό και ωραίο θα ήταν να ενδιαφεραθούμε και για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων του ανθρώπου και σε άλλες χώρες επιτέλους. Ε, ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα ο η Ευρωβουλευτής Αγγέλικα Μλίναρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Ντελαβέντοβα. Δεν κάνουμε λόγο για κάτι καινούριο εδώ και εκπλησόμεθα εδώ όλοι. Από το 2001 γίνονται αυτά τα βασανιστήρια και το 2006 ανακαλύψαμε ότι η CIA ήταν επίσης υπεύθυνη για τις παράνομες κρατήσεις και μεταφορές κρατουμένων στην Ευρώπη πέρα από μια τρομερή παραβίαση δικαιωμάτων του ανθρώπου, πραγματικά δημιουργήθηκε ένας φαύλος κύκλος, δίνοντας στους τρομοκράτες ένα ακόμα επιχείρημα ως πρόσχημα να συνεχίσουν την προπαγάνδα τους και τις τρομοκρατικές τους πράξεις. Τώρα που δημοσιεύτηκε αυτή η έκθεση της Γερουσίας, ήρθε επιτέλους η χρονική στιγμή να δούμε το τι συνέβη στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα κράτη-μέλη δεν είναι καθόλου αθώα όπως αναφέρθηκε από συναδέλφους σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην έκθεση πολλά κράτη γνώριζαν τα γεγονότα αυτής της, αυτών των πράξεων της CIA. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Πολωνία ομολόγησε επιτέλους ότι υπήρξαν αυτά τα γεγονότα και αυτές οι φυλακές. Θα πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση το πρότυπο των ΗΠΑ και να εξετάσει και το επίπεδο συμμετοχής Ευρωπαίων σε όλα αυτά. Πρακτικές για τις οποίες ακούσαμε είναι πραγματικά ανάξιες, απαξιώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν εξεταστικές δράσεις για να δούμε κατά πόσον υπήρξε εμπλοκή σε αυτά τα μέτρα και βασανιστήρια της CIA από πλευράς της Ευρώπης. Ευχαριστώ πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και στην Συνέχεια, από πλευρά Ενωτική Αριστερά, ο κύριο Κώστα Χρυσόγονο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Τι πρακτικέ που χρησιμοποιούσε η CIA επί Προεδρία Μπού για να ανακρίνει κρατουμένου αποτελούν απόδειξη τη έλλειψη πραγματικού σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία διακρίνει τι κυρίαρχε πολιτικέ δυνάμει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Από τη μια παριστάνουν του κίνσορες εκδίδοντας κάθε χρόνο εκθέσεις για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες ενώ από την άλλη οι ίδιοι παραβιάζουν κατάφορα τη σύμβαση κατά των βασανιστήριων που είχαν υπογράψει το. 1994. όμως και η συμπεριφορά της ένωσης ελάχιστα διαφέρει. ενώ η ευρωπαϊκή ένωση διακηρύσσει ότι προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα στην πράξη τα τελευταία χρόνια τα καταπατάει συστηματικά ιδίως τα κοινωνικά δικαιώματα μέσω της επιβολής εξοντωτικών πολιτικών λιτότητας. η μακροχρόνια ανεργία η έλλειψη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης η αδυναμία θέρμανσης σπιτιών το χειμώνα συνιστούν οικονομικά βασανιστήρια. οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποσχέθηκαν στους λαούς τον παράδεισο και σερβίρουν την κόλαση. αλλάξτε πορεία πριν καταστρέψετε την ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε,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 Ο Gianluca Buonanno, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Εγώ θα έλεγα ότι η CIA έκανε καλά αυτά, να κάνει αυτά που έκανε. Ε, υπάρχει φοβερή υποκρισία εδώ πέρα. Όταν ο Ισλαμικός, η Ισλαμική τρομοκρατία κάνει αυτά που έκανε το 2001, σκοτώντας χιλιάδες ανθρώπου, ανθρώπους όπως έκανε στο Πακιστάν τις προάλλες, όπως έκανε στην Αυστραλία. Μα πού ζούμε. Ε, τα βασανιστήρια θα πρέπει να υπάρχουν, τόσο ώστε να ησυχάσει τέλος πάντων και η Ευρώπη κάποια στιγμή. Γιατί αυτοί που είναι τρομοκράτες είναι κτίνοι. Αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα είναι κτίνοι. Και θα πρέπει να μείνει τον Κουαντάναμο ανοιχτό. Τι θα πρέπει να κάνουμε για αυτούς που ε, κόβουν το λαιμό ανθρώπων, που σφάζουν ε, τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας. Ε, στο Ισλάμ υπάρχουν απίστευτες επιταγές. Εμείς αυτή την λογική του μίσου την αλλάξαμε 2.000 χρόνια πριν με τον Χριστό. Η Ισλαμική θρησκεία είναι βία. Ο Νετανιάχου είπε σήμερα ότι η Ευρώπη είναι υποκριτική. Είμαστε υποκριτές. Υποκριτές με όλα αυτά που λέμε για την Παλαιστίνη. Ε, Υπάρχει μια μπλε κάρτα από την κυρία Σπινέλη. Τη δέχεστε? Συνάδελφε, συνειδητοποιείτε ότι με τα λόγια σας επιτεθήκατε έμεσα σε μία σειρά από άθρα του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και σε μία σειρά από θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα εδώ. Σε αυτό το κοινοβούλιο, στο κοινοβούλιο των Ευρωπαίων Δημοκρατιών, έχουμε τοποθετηθεί κατά ε, των βασανιστήριων. Ακόμα και ο δολοφόνο δεν μπορούμε να τον ονομάσουμε κτίνος. Συνα... Συνάδελφε, συνειδητοποιείτε τι λέτε. Φυσικά. Υποκριτικά είναι τα χειροκροτήματά σα. Έρχεται εδώ, έρχεστε εδώ πέρα, κάθεστε στη ζεστούλα σα και δεν πάτε εκεί πέρα να πολεμήσετε υπέρ τη δημοκρατία. Εγώ λέω ότι όποιο έκανε τέτοια σοβαρά αδικήματα δεν μπορεί να θεωρήσει ότι θα πρέπει να προσφέρουμε χαβιάρι και σαμπάνια. Φυσικά, για να καταπολεμήσουμε ορισμένα πράγματα απαράδεκτα, θα πρέπει να κάνουμε και συγκεκριμένε πράξει. Αλλιώ, την τρομοκρατία την αφήσουμε έτσι ξέφραγο αμπέλι. Και στην, τρομο, και στην Ιταλία είχαμε ε, τρομοκρατία. Πώ την καταπολεμήσαμε, Με φυλάκιση, ναι. Αλλά και με αυτού οι οποίοι σφύριζαν πράγματα στου αστυνομικού. Που άνοιγαν το στόμα του. Για ακόμα πιο σοβαρά πράγματα από αυτά που έγιναν στην Ιταλία, ε, εγώ τι λέω, ότι οι Αμερικάνοι μια χαρά τα κάνανε, πολύ καλά κάνανε. Και για να καταπολεμήσουμε την ε, Ισλαμική τρομοκρατία επιτρέπονται τα πάντα. Αυτό που θέλουμε είναι να την νικήσουμε, τίποτα άλλο. Συνέχεια κύριος Κάρλος Κοέλιο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Το 2006 και 2007 αυτό το Ευρωκοινοβούλιο διερεύνησε αυτά τα θέματα μέσω μιας εξεταστικής επιτροπής που είχα την τιμή να προεδρεύω σε αυτήν εγώ. Κάποιοι ισχυρίστηκαν τότε ότι δεν ήταν δυνατόν ένα κράτος δικαίου όπως η ΕΠΑ να έχουν διαπράξει τέτοιες παράνομες πράξεις ε, όπως είχε αναφερθεί. Οι αρχές των ΕΠΑ δήλωσαν ότι αυτές οι κατηγορίες ήταν ασύστατες. Έλεγαν ψέματα όμως. Το Σεπτέμβριο 2006 είχαμε μια μαρτυρία που δεν είχαμε ζητήσει. Ο ίδιος ο George W. Bush, τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, επιβεβαίωσε ενώπιον της κοινή γνώμης ότι υπήρξε αυτό το σύστημα, αυτό το πρόγραμμα και αναγνώρισε ότι είχαν γίνει αυτές οι πράξεις και σε σχέση τώρα με την ύπαρξη των ε, μυστικών φυλακών, τα αναγνώρισε και τις μεταφορές κρατουμένων, όμως αρνήθηκε ότι είχαν γίνει βασανιστήρια. Είπε για άλλη μια φορά ψέματα όμως, όπως απέδειξε η έκθεση της Γερουσίας. Και τέσσερα μηνύματα στέλνει αυτή η έκθεση της Γερουσίας. Πρώτον, Πρέπει να έχει θάρρο για να έχει ηθικό ανάστημα. <clears throat> Όπω η γερουσιαστή Φάινστάιν τόνισε και πολύ σωστά, μόνο ένα όριμο δημοκρατικό κράτο είναι σε θέση να επανορθώσει τα ίδια του τα λάθη και να συνεισφέρει ώστε να αποκλειστούν αυτά στο μέλλον. Δεύτερον, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τι προσπάθειε να αποκαλυφθεί και να λάμψει η αλήθεια. Χωρί τι προσπάθειε αυτέ δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι θα αποκαλυφθεί η αλήθεια. Ιδιαίτερα όταν οι εθνικέ κυβερνήσει δημιουργούν διαρκώ εμπόδια για την αποκάλυψη τη αλήθεια. Επαναλαμβάνω αυτό που πολλέ φορέ επανέλαβα σε αυτό το ημικύκλιο είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δεχθούμε, να επιβάλλεται δηλαδή το κρατικό απόρριτο στην αλήθεια και στα θεμελιώδη δικαιώματα και πρέπει να συνεισφέρουμε στην αποκάλυψη αυτών των θεμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίτον, ο σκοπό όποιο και αν είναι ποτέ δεν δικαιολογεί τα μέσα. Δεν μπορούμε να δεχθούμε τα βασανιστήρια. Καταδικάζονται από το διεθνέ δίκαιο και όπω αποδεικνύεται εδώ δεν είναι δυνατό να, να ε, συμβαίνουν. Το αποδεικνύει και η έκθεση τη Γερουσία. Επίση διαπιστώνεται ότι υπάρχει έλλειμμα, τέταρτο αυτό, στον δημοκρατικό έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών. Δεν λειτουργήσε αυτό ο έλεγχο, ε, ο δημοκρατικό έλεγχο. Και η CIA έλεγε διαρκώ ψέματα. Έχουμε το ίδιο πρόβλημα όμω και στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και στην συνέχεια δέχεστε ε, μπλε κάρτες. Έχετε μια μπλε κάρτα. Την δέχεστε παρακαλώ. Thank you. Um, agree with what's being said in here. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με όσα λέγονται εδώ συμφωνείτε στο ότι δεν έχει νόημα οι εξεταστικές επιτροπές τελικά να καταλήξουν σε πορίσματα τα οποία το μόνο που θα κάνουν είναι να βρίσκουν από διοποδέους τράγους τον εκάστοτε ανακριτή ενώ θα αφήνουν ταυτόχρονα ελεύθερους τους πολιτικούς που διέταξαν τέτοιου είδους βασανιστήρια. Συμφωνείτε με αυτό παρακαλώ. Σίγουρα συμφωνώ μαζί σας γι' αυτό. Για την έκθεση η αξία δεν είναι μόνο ο επιμερισμό ευθυνών. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Αλλά όπως πολύ σωστά αναφέρθηκε πρέπει να διακριβωθούν οι ευθύνες όλων. Εκείνων που ενέκριναν, εκείνων που διέπραξαν. Ωστόσο κυρίως η αξία τη της διακρύβωσης είναι το να μάθουμε και να μην επαναλάβουμε τα ίδια λάθη στο μέλλον. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Στη συνέχεια, Βάιντεν Χόλτσερ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Η ελευθερία είναι τα θεμέλια της δυτικής ε, κοινωνίας των κοινότητας των εθνών και η προστασία αυτών των δικαιωμάτων είναι έργο όλων μας. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι σε κάποιες καταστάσεις και υπό κάποιους όρους και προϋποθέσεις και περιορισμοί αυτών των δικαιωμάτων μπορεί να απαιτούνται. Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν μια τέτοια κατάσταση και πολλά από αυτά τα μέτρα σε σχέση με τα όσα συνέβησαν ε, ήταν υπερβολικά και συνέβησαν και προκλήθηκαν από αυτό το γεγονός και επιβεβαιώνονται αυτά μέσω της έκθεσης CIA και για την πολιτική ασφάλειας πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος έλεγχος μεγαλύτερη εποπτεία γιατί διαφορετικά θα υπάρχει διαρκώς μεγαλύτερη ε, καταπίεση με μικρή επιτυχία όλα αυτά τα βασανιστήρια. Η απειλή των τρομοκρατών αυξήθηκε από τότε. Σε ένα γερμανικό περιοδικό λέγεται ότι ήταν ο μεγαλύτερος θρίαμβος του Οσάμα Μπιν Λάντεν που μπόρεσε να αποδείξει ότι είναι ένα κράτος που παρανομεί η ΕΠΑ. Πρέπει να πούμε με την προσθήκη ότι η επεξεργασία αυτών των ε, παράνομων γεγονότων με εντυπωσιακό τρόπο ολοκληρώνεται από τη Γερουσία και αποδεικνύεται ότι οι ΕΠΑ θέλουν να είναι και είναι κράτος δικαίου. Είναι σημαντικό στοιχείο αυτό. Δεν πρέπει όμως αυτό να μας οδηγήσει σε αυταρέσκεια και να είμαστε ικανοποιημένοι. Πρέπει να επεξεργαστούμε και να αναλύσουμε αυτά τα τρομακτικά στοιχεία, ιδιαίτερα όσον αφορά τον ρόλο επιμέρους κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποινικέ πράξεις που πρέπει ως ποινικέ πράξεις να διώκονται και δικαστικά να καταδικαστούν και να ε, υποστούν οι αρμόδιοι υπεύθυνοι τις συνθήκες. Αυτό είναι το μήνυμα που μας δίνει αυτή η έκθεση. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε πολύ. Και στη συνέχεια τώρα θα λάβει τον λόγο ο κύριος Τζαμπάσκι, ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναμφίβολα η αποκάλυψη αυτών των συμβάντων στην έκθεση της Αμερικανικής Γερουσίας όσον αφορά στις απαγωγές και στην κακομεταχείριση των κρατουμένων δείχνει ότι η χώρα η οποία ε, διεκδικεί για τον εαυτό της το δικαίωμα να προστατεύει περισσότερο από οποια οποιασδήποτε άλλες χώρες τα δικαιώματα των πολιτών ε, ε, δεν ανταποκρίνεται στο το οποίο λέει. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ε, δεν μπορεί κανείς να προβάλλει τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας για να δικαιολογεί αυτή της πράξης και οι κατασυρωοί δολοφόνοι το ίδιο που θα μπορούσαν να πούν. Νομίζω ότι χρειάζεται να ασκηθούν ποινικέ διώξει για αυτέ τι παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνού δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Βάιγκελ από τους φιλελεύθερους για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εισαγωγικά θα ήθελα να σας πω ότι είμαι ικανοποιημένος με τη σημερινή σας ομιλία και την αξιολόγηση που κάνατε. Θα ήθελα να πω όμως ότι όταν βλέπουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις, όταν τις είδαμε στους Δήμους Πύργους, εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Εξακολουθεί να ισχύει αυτή η αλληλεγγύη. Δηλαδή, Δυστυχώ, ο λεγόμενος πόλεμος για την τρομοκρατία τα επόμενα χρόνια δημιούργησε μία σειρά από σοβαρότατα ερωτήματα. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε το γεγονός ότι οι ΕΠΑ κατέστρεψαν τη φήμη ευρωπαϊκών κρατών που ήταν σύμμαχοι με τη ΗΠΑ. Οι Αμερικάνοι είναι ο, η μία χώρα από τις 165 που έχουν προσυπογράψει τις διεθνείς συμβάσεις και θα πρέπει να διώξουν τους ένοχους. Αν οι Αμερικανοί αποφασίσουν να μην κάνουν τίποτα και να μην τιμωρήσουν τους υπεύθυνου. μπορεί να υποστούν την ρήτρα του ICC, του ποινικού δικαστηρίου, που έχει τη δυνατότητα να δράσει αυτεπάγγελτα όταν η ίδια η χώρα δεν δρά εναντίον των ενόχων της. Μπορεί να εκδώσει δηλαδή ένταλμα σύλληψης εναντίον όλων των ενόχων και να τους διώξει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έκαναν πάρα πολύ λίγα πράγματα. Έκαναν μόνο το πρώτο τμήμα στην προσπάθεια αποκάλυψης ε, της αλήθειας και έχω αναλάβει μόνο ένα μικρό τμήμα των δεσμεύσεων. Αλλά μην ξεχνάτε ε, ότι το μου είναι ακόμα ανοιχτό. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Παύλο Ιγκλέσιας από την ΚΟΕ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το να, να βάλει κανεί τρόφιμα και αντικείμενο στο ορθό του κρατούμενο, να χύνει υγρά στα γενετικά όργανα του κρατούμενου, να τον αφήνει επί μέρε ε, ολόκληρε χωρί ύπνο, να τον απειλεί ότι θα ασκήσει βία στη μητέρα του, να τον απειλεί ότι θα τον αφήσει ανάπηρο. Αυτέ είναι οι πρακτικέ που μάθαμε διαβάζοντα την έκθεση αυτή. Το πρόβλημα δεν είναι ότι ανθρώπινα όντα ήταν ικανά να διαπράξουν τέτοιου είδου φρικαλαιώδει πράξει σε άλλα ανθρώπινα όντα, γιατί πάντοτε θα υπάρχουν τέτοια ανθρώπινα όντα. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν φασίστε βουλευτέ που υπερασπίζονται τα βασανιστήρια σε αυτή την αίθουσα, οι οποίοι φορούν γραβάτα και κουστούμι. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτήν εδώ την αίθουσα τολμούν ε, βουλευτέ να επικαλούνται και να στηρίζουν τέτοιου είδου πρακτικέ. Συμμετείχαν τέτοιου είδου βουλευτέ σε κυβερνήσει που συνεργάστηκαν με τη CIA. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόρδιν Νίκε για 1,5 λεπτό από τους μη εγγεγραμμένους. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπροκ, ο κύριος Ιγκλέσιας έχουν απόλυτο άδικο. Η δημοκρατία είναι η τυραννία των πολλών. Η πλειοψηφία δεν ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θέλει την ασφάλεια ό,τι και να κάνουμε, βασανιστήρια, κακομεταχείριση κτλ. όλα παίζουν. Ε, για την Πολωνία αυτή η Εξεταστική Επιτροπή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Η πολωνική κυβέρνηση τα αρνήθηκε όλα καταρχήν. Υπάρχουν άτομα τα οποία αρνήθηκαν την ύπαρξη βασανιστήριων στην, ε, και την άσκηση βασανιστήριων στην Πολωνία. Ο Πρωθυπουργό της Πολωνίας, που ήταν επικεφαλής των διαπραγματεύσεων για τις συνθήκες ε, Ένταξη τη Πολωνίας είναι αυτός ο οποίος ήρθε σε επαφή με τη CIA. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά για το θέμα, αλλά δεν έχω χρόνο αυτή τη στιγμή. Σας ε, συνιστώ να ασχοληθείτε περισσότερο με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Ντανιέλ Μπούντα από το ΕΛΚΑ για δύο λεπτά ευχαριστώ. η απόπειρα στις 11 ε, ε, Σεπτεμβρίου, οι επιθέσεις της Μαδρίτης, του Λονδίνου, της Βοστόνης δείχνουν ότι καμία χώρα δεν είναι στο απειρόβλητο και μπορεί να υποστεί ε, φοβέρε φοβερές επιθέσεις και να χαθούν χιλιάδε ζωέ. Ε, όλα αυτά εντυπωσίασαν όλο τον κόσμο, όχι τις Ηνωμένες και αποφασίσαμε από κοινού να προσπαθήσουμε να γίνουμε επιθετικοί αντί για αμυντικοί. Σήμερα το Ισλαμικό κράτος ε, κάνει στρατολογή κόσμο και ε, εξαιτία τη πόλωσης της κοινωνίας βρίσκει όλο και περισσότερους. οι αξίες μας κινδυνεύουν. Αθώοι κάθε μέρα είναι θύματα της τρομοκρατίας, μια άθλιας τρομοκρατίας. Και τα θύματα αυτά δείχνουν ότι η απειλή της τρομοκρατίας είναι πραγματικότητα. Οι άνθρωποι αυτοί συχνά που είναι ε, οι θήτες έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια. Η τρομοκρατία δεν έχει σύνορα. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι αιτίε της τρομοκρατίας και να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε βασικά ερωτήματα. Τι πρέπει να κάνουμε, ούτως ώστε αυτό το φαινόμενο να μειωθεί. Να γι' αυτό η υπερβολική πολιτικοποίηση του φαινομένου δεν βοηθάει κανένα. Τούτου λεχθέντος ποτέ δεν θα δεχτούμε να χρησιμοποιηθούν απάνθρωπες μεθόδους για να πάρουμε πληροφορίες. Θα πρέπει να σταματήσει η απάνθρωπη συμπεριφορά, θα πρέπει να σταματήσουν τα, βασανιστήρια. Αλλιώς τα θύματα γίνονται θύτες κάποια στιγμή. Ο κοινό στόχος όλων των εθνών θα πρέπει να είναι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας όπου και αν βρίσκονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Άννα τώρα εκ μέρους των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Η έκθεση της Γερουσίας επιβεβαιώνει αυτό που και, τα, και οι εκθέσεις του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχουν αντοπίσει από το 2007. Όμως προσθέτει νέες λεπτομέρειες οι οποίες είναι ατριχιαστικές και για τα βασανιστήρια και για τα άλλα εγκλήματα της CIA, για τις ε, συλλήψεις των τρομοκρατών και για τις μυστικές φυλακές που ε, φαίνεται ότι έχουν δώσει σε υπεργολαβία σε υπαλλήλου με πρόσχημα τον Καντάφη και τον Μουμπάρακ και επίσης τις, κυβέρ... τις πράξεις της κυβέρνησης Μπούς ε, που δείχνουν την αμερικανική ε, προσέγγιση του θέματος διεθνώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Γερουσία ήδη με πέντε ε, χώρες από αυτό το κοινοβούλιο είχε επιτρέψει τη συνεργασία με τη CIA και με την εξαγωγή ε, κρατουμένων ε, επιβεβαιώνεται η έπραξη μυστικών φυλακών στην Ευρώπη όπως τη Λιθουανία και την Πολωνία με τη συνενοχή ε, των χωρών αυτών. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωκοινοβούλιο να εξεύρει ένα μηχανισμό διερεύνησης και εξέτασης των όσων έχουν συμβεί στα πλαίσια αυτής της πολιτικής των ΗΠΑ που δεν μπορούν να παραμένουν στην ατιμορρησία. Η χώρα η Πορτογαλία είχε κάνει μια, μερικές από τις πρώτες πτήσεις ε, ε προς τον Κουαντάναμο μετά τις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Και το 2006 και 2007 πάνω από 100 φορές υπήρξαν διελεύσεις από το πορτογαλικό έδαφος ε, με την ε, ε, συνενοχή των πορτογαλικών αρχών ήταν αναρμόδιες και ανίκανες πορτογαλικές αρχές για να ε, εμποδίσουν αυτές τις ενέργειες αλλά αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί. Ήταν απλώς ε, ανίδες ή συνένοχες. Η χρήση επίσης της βάσης της Αζόρες αξιοποιήθηκε και η χώρα μου με επονίδιστα από το 2007 αποκρύπτει την αλήθεια, εμποδίζει την έρευνα των μυστικών υπηρεσιών και τη δικαστική έρευνα και θα πρέπει να ε, δώσει στο Ευρωκοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια τι πτήσει που επιτράπηκαν προ το Γκουαντάναμο με μια εξεταστική επιτροπή που θα πρέπει να δημιουργηθεί σε αυτό το Κοινοβούλιο. Κυρίε και κύριοι, πόσε φορέ δεν θα πρέπει να σκεφτούμε ότι τι δικέ μα τι ευθύνε πρέπει να τι αναλαμβάνουμε οι ίδιοι, να μην τι επιρρύπτουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που παρόλα αυτά είχε ω επικεφαλή τον ε, πρώην ε, Πορτογάλο Πρωθυπουργό, τον Μανουέλ Ζωζέ Μπαρόζο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα για όλου μα, για την Πορτογαλία και για όλη την Ευρώπη. Ευχαριστούμε. Γαλάζια κάρτα. Τη δέχεστε. Ε, ερώτηση από τον κύριο Μαρίνιο. Ο κύριος Μαρίνιο. Ευχαριστώ. Κυρία Γκόμες, αγαπητή συνάδελφοι. Ακούμε πολλά δημόσια, πολλές δημόσιες τοποθετήσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους φορέων που δημιουργούν τοπέδα συγκέντρωσης όπως το Γκουαντάναμο ή που επιτρέπουν στους εαυτούς τους να διαπράττουν βασανιστήρια όπως αυτά που τώρα καταγγελθήκαν από την Αμερικανική Γερουσία. Πιστεύετε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που επέτρεψαν τα βασανιστήρια της CIA στην επικράτειά τους θα πρέπει να τιμωρηθούν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. οι μεγάλες δημοκρατίες πρέπει να αποδέχονται τα σφάλματά τους. Αυτό συνέβη με την Αμερικανική Γερουσία. Αλλά αυτό ήδη ζητά το Ευρωκοινοβούλιο και γι' αυτό αυτή τη στιγμή θα πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά μας. Να φροντίσουμε να βρούμε τους ε, Ευρωπαίους υπετίους και να μην αφήσουμε ατιμόρυτα τα εγκλήματα ενώπιον όλων. Θα πρέπει να αναλυθεί δράση για όσους ε, έδωσαν τις εντολές για αυτές τις βάρβαρες πράξεις που ε, διαπράχθηκαν από τη CIA με τη συνενοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Τώρα ο κύριος Φωνστόρχ, η κυρία Φωνστόρχ, ε, ένα λεπτό, από τις 6.000 σελίδες, μόνο 500 σελίδες έγιναν γνωστές, δημοσιεύθηκαν και διαπιστώνουμε ότι έχουν γίνει βασανιστήρια ανεξέλεγκτα. Τα βασανιστήρια ούτως ή άλλως πρέπει να είναι απόλυτα απαράδεκτα. Η διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λέει ότι κανείς δεν θα πρέπει να υπόκειται σε βασανιστήρια. Διαπιστώνω πρώτον τα βασανιστήρια είναι μεσαιωνικέ μέθοδοι ή μέθοδοι κρατών όπου δεν υπάρχει δίκαιο. Όχι κρατών του 21ου αιώνα. Δεύτερον, όποιος βασανίζει πρέπει να τιμωρείται. Οι υπέτη πρέπει να τιμωρηθούν από τα εθνικά ή τα διεθνή δικαστήρια και γι' αυτό είναι επιτέλους χρόνος οι Ηνωμένε Πολιτείε να αναγνωρίσουν το Διεθνές ε, Ποινικό Δικαστήριο και να μην προστατεύουν τους υπετίους και τους βασανιστές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος ε, Χαβιέ Κόσο Περνόη. Ένα λεπτό. Οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται έχουν περάσει σε φοβερές λεπτομέρειες. Βασανισμοί, βασανισμοί, βασανισμοί. Ένα είναι το κοινό. Πρέπει να το επαναλαμβάνουμε αυτό συνέχεια είναι οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2012 είχαμε ένα ψήφισμα που έλεγε να ερευνήσουμε τις επιπτώσεις του προγράμματο αυτού και τη συμμετοχή των χωρών μελών. Ντρέπομαι που ξέρω ότι η χώρα μου συνεργάστηκε στα βασανιστήρια αυτά και στις απαγωγές ανθρώπων, όπως ε, έγινε και με τις μυστικές ε, φυλακές στη Ρουμανία, τη Λιθουανία και αλλού όπου συνεργάστηκαν πολλές χώρες μέρη. Το ψήφισμα πρέπει να ζητάει την καταδίκη και να ζητάει πάνω απ' όλα έρευνα, προκειμένου να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, οι όσοι συνεργάστηκαν και να πάνε στη δικαιοσύνη. Να καταδικαστούν να μην επαναληφθούν τα ίδια φαινόμενα. Αλλιώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να δικαιούται να μιλάει για ανθρώπινα δικαιώματα πια. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Ένα λεπτό, Ζιλ Breton. Η έκθεση που μόλις δημοσιεύτηκε αποκαλύπτει ότι η CIA για χρόνια μετέρχεται βασανιστήρια. Αυτό δεν μας εκπλήσει. Πολλά παραδείγματα αποδεικνύουν ότι οι ΗΠΑ έχουν γίνει μια επιθετική δύναμη και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με δυσπιστία. Το σκάνδαλο Wikileaks μας έμαθε το 2013 ότι η NSA έκανε κατασκοπία μεγάλης κλίμακας ακόμη και εναντίον ε, συμμάχων και πολιτικών τους όπως η Φρανσουά Λάντ και η Άγγελα Μέρκελ. Το 1796 το, συγγνώμη, το 1996 το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε παράνομα μέτρα. Το 2014 οι Ηνωμένε Πολιτείε επέβαλαν 6,5 δις ε, πρόστιμο σε μια γαλλική τράπεζα BNP επειδή συνεργάστηκε με κράτη που είναι στην μαύρη λίστα της. Και ήδη όμως το 2014 αποσταθεροποίησαν ηθελημένα την Ουκρανία, προκαλώντας κίνδυνο πολέμου με, την Ουκρανία, με τη Ρωσία. Πόσες ε, περαιτέρω ταπεινώσεις και προκλήσεις θα ανεχθεί η Ένωση πριν καταλάβει ότι πρέπει να αντιδράσει αρνούμενη να υπογράψει την σύμβαση TTIP. Ευχαριστώ, όλοι ο Πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος Τσάμπα Σόγκο από το ΕΛΚ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Οπωσδήποτε. Είναι σημαντικό το ότι λάβαμε πληροφόρηση για το ότι αυτά που γίνονται είναι απόλυτα απαράδεκτα. Για μένα αυτές οι πρακτικές της CIA είναι αποτρόπαια. Αποτρόπες, ακόμη και αν ε, ε, ορισμένοι το υποστηρίζουν και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι και σε άλλες χώρες έχουν γίνει αυτά και με ανησυχεί ιδιαίτερα ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί και ε, από τις ΗΠΑ. Όταν τίθενται ε, εν κινδύνο τα συμφέροντά τους δεν παίζουν κανένα ρόλο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η δικαιοσύνη δεν καταφέρνει πάντα να συμβαδίσει με τα εγκλήματα αλλά η δικαιοσύνη είναι τμήμα αυτών που διαχωρίζουν ε, τα κράτη δικαίου από τα υπόλοιπα. Εάν εμείς δεν τηρούμε τις προδιαγραφές που εμείς αποφασίσαμε, δεν έχουμε μάθει τίποτα από την ιστορία του 20ου ε, αιώνα. Ευχαριστώ. Τώρα η Κάτι Πύρη. Από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, δύο λεπτά. Πρόεδρε, η έκθεση της Αμερικανικής Γερουσίας δείχνει τα βασανιστήρια και το μέγεθος βασανιστήριων που έλαβαν χώρα μετά την 10η Σεπτεμβρίου. Τώρα πια έχει αποδειχτεί, παρόλο που υπήρχαν υπένιες όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε μάθει πολλά και έχουμε μάθει και ότι η σεπτεμβριου τωρα πια εχει αποδειχτει παρολο που υπηρχαν οι συμμετείχε και παρόλα αυτά η Ευρώπη δεν λέει τίποτα και ούτε είναι απόλυτα ρητό το ψήφισμά μας. Οι χώρε μέλη από ό,τι φαίνεται συνεργάστηκαν στι πρακτικές αυτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Συμβούλιο της Ευρώπης έπαιξε ένα σημαντικό ρολό πριν από μερικά χρόνια όταν έπαιξε τις αποδείξει και δεν άφησε να φανεί η συμμετοχή κυβερνήσεων στις παράνομες απαγωγές, ότι χρησιμοποιήθηκαν αεροδρόμια, αεροπλάνα ή ακόμα και ότι υπήρχαν σε ευρωπαϊκή επικράτεια Φυλακέ. Πρόκειται για παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και είναι κάτι πολύ βασικό αυτό για τι δικέ μα αξίε, τι ευρωπαϊκέ αξίε. Εμεί θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη δρομοκρατία, αλλά δεν είναι δυνατόν να παραβιάζουμε συγχρόνω τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η έκθεση αυτή λοιπόν τη Αμερικανική κυβέρνηση πρέπει να ληφθεί υπόψη και να αποτελέσει ένα μάθημα για μα για το μέλλον. Είναι πολύ βασικό προκειμένου οι χώρε μέλη να αναρωτηθούν δεν ήρθε πια η ώρα να δουλέψουμε κι εμείς για αυτά τα θέματα για να καταδικάσουμε αυτές τις πρακτικές. Είναι πολύ βασικό για την ίδια την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να είναι στην πρώτη γραμμή των ανθρωπένων δικαιωμάτων. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια ε, μαύρη σελίδα στην ιστορία μας. Ζητάμε λοιπόν και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει έρευνες για τις παρεβιάσεις του διεθνούς δικαίου που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό έδαφος και να συνεργαστούμε με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των ΗΠΑ. Είναι πράγματα που πρέπει να προχωρήσουν γιατί τελείως θα μας κυνηγάνε διαβίου. Συνεπώς, Πρόεδρε, πρέπει να φροντίσουμε να ζητήσουμε και τις ευθύνε των κυβερνήσεων που αναμίχθηκαν σε τέτοιες πρακτικές. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κλούνε. Δύο λεπτά. Ο ε, κύριε Κλούνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η... Το σκοτεινό πέπλο που καλύπτει πλέον την εικόνα των ΗΠΑ με τις μυστικές υπηρεσίες να θέτουν ένα αμφιβόλο την ασφάλεια, την ασφάλεια των πολιτών όλου του κόσμου, με τον ίδιο τον πρόεδρο Ομπάμα ε, να αναμειγνύεται εδώ γύρονται πολλά ερωτήματα για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλές από τις ε, χώρες μέλη. Μιλάμε για βασανιστήρια και την ε, παραβίαση των θεμελιωδέστερων αξιών και έτσι δίνουμε δικαιώματα στους εξτρεμιστές που αυτό ακριβώς αναζητούν το να δρά κατά των αξιών που προασπίζεται είναι αντιπαραγωγικό Και βεβαίως δίνει κάθε δικαιολογία στις ε, ομάδες αυτές της τρομοκρατίας να συνεχίζουν τη δική τους ε, τακτική. Με τον αποκεφαλισμό ε, των εργαζομένων σε μη κυβερνητικέ οργανώσεις, των εργαζομένων σε φιλανθρωπικές, σε φιλανθρωπικές ομάδες, εμείς δεν μπορούμε να κρατήσουμε την ίδια στάση όταν δεν έχουμε σεβαστεί αυτές τις αξίες. Η έκθεση αποδεικνύει ότι φυλακισμένοι άντρες και γυναίκες βασανίστηκαν σε, επίπεδο που έφτασαν να έχουν πρόβλημα με την υγεία τους. Βεβαίως κάποιοι ευαγγελίζονται ότι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Όμως οι δημοσκοπήσεις λένε ότι 51% των Αμερικανών δέχονται τα βασανιστήρια της CIA ως δικαιολογημένα διότι έτσι προλήφθηκαν τρομοκρατικές επιθέσεις. Η Σύμβαση της Γενέβης και του ΟΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι συμβάσεις κατά των βασανιστήριων, οι συμβάσεις αυτές έχουν κυρωθεί σχεδόν από όλες τις χώρες του κόσμου συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ. Δεν μπορούμε λοιπόν να επιτρέψουμε τα πρότυπα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε στιγμές ε, σύγκρουσης να παραβιάζονται τελείως. Και δεν μπορούμε να πέφτουμε στο χαμηλότατο επίπεδο των τρομοκρατικών οργανώσεων. Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη με αφορμή αυτή την έκθεση. Τα δικαστήρια να ε, δώσουν τη συνέχεια που αρμόζει στα πορίσματα της έκθεσης αυτής. Και τώρα η Σιλβή Φων δύο λεπτά παρακαλώ. Οι απαγωγές, οι εξαφανίσεις, ε, η έλλειψη ύπνου, ο περιορισμός σε μικρά κουτιά, το waterboarding, είναι μακρύς ο κατάλογος των βασανιστήριων και είναι πραγματικά αποτρόπαιος. Και γι' αυτό δεν μπορούμε παρά να χειροκροτήσουμε την πρόεδρο της Επιτροπής Έρευνας τη Αμερικανική Γερουσία. Αλλά από τις 6.000 σελίδες της μυστικής έκθεσης, μόνο 500 δημοσιεύθηκαν. Και ένα μεγάλο τμήμα των σελίδων που δημοσιεύθηκαν είναι διαγραμμένες. Αυτό σημαίνει ότι όλα μπορούν να συμβούν και τα περισσότερα που έχουν συμβεί είναι ακόμη ε, μυστικά. Η Επιτροπή, η αντίστοιχη της ε, Αμερικανικής Βουλής ήδη από το 2006 είχε ερευνήσει αυτό το θέμα και είχε ζητήσει να υπάρξει πλήρης διερεύνηση. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Κανένα σκοπός δεν είναι δυνατόν να δικαιολογήσει αυτά τα φρικαλαία μέτρα, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η CIA που είναι κατάφορη παραβίαση των αρχών μας. Αλλά το να καταδείξουμε ως ενόχους μόνο τις ΗΠΑ δεν αρκεί. Κάποιοι για λόγους πίστης προς τις συμφωνίες που έχουμε τις ΗΠΑ ή για λόγους ε, χρηματικής αμοιβή συμμετείχαν και αυτοί και πρέπει και αυτοί να ελεγχθούν. Αυτό είναι καθήκον που έχουμε προς τα θύματα και προς τη δική μας εξοπιστία. Ο πρόεδρος Βασνεύσκη και ο, ε, ο, επικεφαλής της προηγούμενης, ε, ο προηγούμενος επικεφαλής της Ρουμανικής Μυστικής Υπηρεσίας τώρα μετά την, ε, τις αποκαλύψεις αναγκάστηκαν να παρδεχθούν ότι υπήρχαν μυστικές φυλακές στις χώρες τους και η Βρετανική κυβέρνηση από ό,τι διάβασε στο γερμανικό τύπο πριν τη δημοσίευση της έκθεσης του Σενά, της ε, Γερουσίας είχε πει ότι αναφορές για βρετανική συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό πρέπει, είχε ζητήσει να μην γίνει δημόσια. Αυτές οι στρατηγικές ε, παραπλάνεις των κυβερνήσεων πρέπει να σταματήσουν. Όλα τα κράτη της Ένωσης έχουν υπογράψει τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το άρθρο 3 λέει ότι κανείς δεν πρέπει να υπόκειται σε βασανιστήρια, σε ταπεινωτική μεταχείριση δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε αυτά τα φαινόμενα με ασυδοσία και χωρίς να τα καταγγέλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Και τώρα, από την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού ο κύριος Λέναρτ. Ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή της Αμερικανικής Γερουσίας ε, δείχνει φτυχτά πράγματα τα οποία έκανε η CIA την περίοδο 2001 με 2009 σε κρατούμενους. Τις πρακτικές που χρησιμοποίησε, δεν τους άφηνε να πεθαίνουν, τις πείνας κλπ. κλπ. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν την φρίκη μας απέναντι σε τέτοια βασανιστήρια. Συγχρόνω, βέβαια πολύ σωστά διάφοροι συνάδελφοι είπαν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα το ότι δημοσιοποίησε την έκθεση αυτή η Αμερικανική Γερουσία. Είναι το πρώτο βήμα για διαφάνεια και για προβληματισμό. Προβληματισμό από την πλευρά μας που είναι κάτι πολύ βασικό για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Και θα ήταν καλό αν είχαμε και ολόκληρη την έκθεση της Αμερικανικής Γερουσίας και οι ευρωπαϊκές χώρες από τη δικιά τους την πλευρά να κάνουν τα σωστά βήματα για να υπάρξει διαφάνεια για αυτή την υπόθεση και έτσι η Ευρώπη να μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη. Είναι σημαντικό ότι αναφέρεται το τι έγινε με τους κρατούμενους στην πτέρυγα εκείνη του 119 όπως αναφέρεται στην έκθεση. Τι έχει γίνει όμως με άλλους κρατούμενους από Αφγανιστάν, Ιράκ και τα λοιπά είχαν την ίδια τύχη. Καλό θα ήταν να το ξέρουμε και αυτό. Θα ήταν καλό να είχαμε περισσότερες πληροφορίες και περισσότερη διαφάνεια και για αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε να κάνουμε με άγνωστες συμπεριφορές και είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλειά μας και την ασφάλεια των γειτόνων μας να ξέρουμε περισσότερα. Δεν είναι δυνατόν να παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα και να μην πέφτουμε στη συζήτηση που ίσως θέλουν να κάνουν μένες πολιτείες και ο Τσένι όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των βασανισμών. Τα βασανιστήρια είναι απαράδεκτα. Τελεία και παύλα. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα η Ελένα Βαλενθιάνο. Από τη σωσταστική ομάδα, δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το κοινοβούλιο μας πρέπει να ανοίξει πάλι την Ερευνητική Επιτροπή, η οποία δούλεψε το 2006 και το 2007, προκειμένου να μάθουμε τι ακριβώς έγινε με τις πτήσεις αυτές τη CIA. Γιατί δεν δικαιολογούνται τα μέσα από το σκοπό. Είναι πολύ σημαντικό και ο σκοπό και τα μέσα. Ξέρουμε ότι η Αμερικανική Γερουσία έκανε παραδειγματική δουλειά. Αλλά δεν μπορούμε απλώς να αρκεστούμε στην αναγνώριση αυτής της παραδειγματικής δουλειάς. Το Κοινοβούλιο μας το 2006 και 2007 και ήμουν μέλος της ε, μόνιμης αυτής επιτροπής ερεύνησε την κατάσταση με πάρα πολλές δυσκολίες. Τα προγράμματα δηλαδή αυτά που είχαν πτήσει στη CIA. Η Γερουσία έκανε τη δικά της την έκθεση και πια η δικιά μας η έκθεση δεν έχει νόημα. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξανανοίξει η έρευνα, να ξαναγίνει, να γνωρίζουμε την πραγματικότητα για να καταλογιστούν ευθύνες. Με πολλές δυσκολίες δουλέψαμε την προηγούμενη φορά και το χρωστάμε στους πολίτες οι οποίοι μας παρακολουθούν. Βλέπετε για να μπορούμε να δίνουμε μαθήματα, όπως κάνουμε αυτή τη βδομάδα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Σουδάν, στη Μαυριτανία, στη Βενεζουέλα, στην Αίγυπτο κλπ, πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε σε θέση να αποτελούμε εμείς παράδειγμα. Η σημερινή συζήτηση λοιπόν πρέπει να είναι η αρχή και όχι το τέλος μιας δουλειά που πρέπει να ολοκληρώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που άρχισε το 2006 αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Αυτό ζητούμε λοιπόν από πλευρά των σοσιαλιστών. Θέλουμε να ανοίξει και πάλι η Ερευνητική Επιτροπή. Κρίμα που δεν εδώ ο κύριος Μπροκ. Πρέπει να κλείσει το Γουαντάναμο. Ανεξάρτητα από το αν υποδέχονται οι χώρε του κρατούμενου του Γουαντάναμο ή όχι. Έτσι κι αλλιώ όταν άνοιξαν αυτέ οι φυλακέ δεν μα ρώτησαν τη γνώμη μα. Ευχαριστώ. Catch the Τώρα, λέει ο πρόεδρος και πρώτος είναι από το ΕΛΚ, ο Μίχαλ Μπόνι. Παρακαλώ. Η δικαιοσύνη ως ειρήνη και ελευθερία είναι η βάση των αρχών μας και δεν αφήνει περιθώριο για βασανιστήρια. Πρέπει να εξετάσουμε υπεύθυνα τα μέσα που χρησιμοποίησε η CIA και να αποτιμήσουμε τις επιπτώσεις. Οι πολωνικές αρχές το 2008 έδωσαν τη δυνατότητα στη CIA να συλλάβει και να κρατήσει σε φυλακές ορισμένους υπόκτους αλλά όχι να τους βασανίσει. Οι αρχές εκείνη την ε, περίοδο ζήτησαν ένα ειδικό υπόμνημα για τους κανόνες λειτουργίας αυτών των φυλακών αλλά δεν τους εστάλησαν αυτοί οι κανόνες. Το 2009 υπογράψαμε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες επί κάποιων κανόνων ιδιαίτερα για το να υπάρχει πολωνική δικαιοδοσία για τους Αμερικανούς αξιωματικούς που εργάζονται στην Πολωνία. Η πολωνική εισαγγελία εξετάζει το θέμα αυτό. Η έκθεση της Αμερικανικής Γερουσίας είναι εσωτερικό θέμα και καθήκον των Αμερικανικών αρχών. Αλλά οι απαντήσεις στις ερωτήσεις εάν στη χώρα μου έγιναν βασανιστήρια είναι θέμα της δικής μου χώρας. Ωστόσο πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας. Σε οποιαδήποτε χώρα μπορεί να προκύψει αυτό το πρόβλημα, πώς να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των πολιτών Αποφεύγοντας όμως ε, τη χρήση τέτοιων αποτρόπαιων μέσων, ενώ έχουμε βέβαια την υποχρέωση να αντιμετωπίσουμε τους πραγματικούς κινδύνους, που, τους κινδύνους όπως είναι η τρομοκρατία, ε, λαμβάνοντας υπόψη και τι συνέβη τις τελευταίες δύο μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Από πλευρά των Σοσιαλιστών, ο Νίκολα Καπούτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η πρόσφατη έρευνα τη ε, έκθεση τη Γερουσία για τα βασανιστήρια τη CIA δείχνει την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι δραματικά τα στοιχεία αυτά, γιατί φαίνεται ότι πρόκειται και για ένα πρόγραμμα που ακόμα και από τον πρόεδρο Ομπάμα έχει εγκριθεί. Με εικονικό πνιγμό, με άλλε μορφέ βασανιστήριων, με τον απόλυτο έλεγχο και την ε, πλήρη εξοπαίδωση των κρατουμένων φαίνεται ότι δεν μπορεί οι πληροφορίες αυτές να αποσπώνται με όποιον ε, τρόπο γίνεται. Αυτά βέβαια θεωρούνται μέρος του παρελθόντος, αλλά δεν είναι έτσι. Αν θέλουμε να είμαστε πολιτισμένες χώρες θα πρέπει να καταδικάσουμε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Δεν ε, αρκεί να Μάλλον αυτή, αυτός ο εξευτελισμός του ανθρωπίνου όντως είναι ένα σκόλαφος και για οποιαδήποτε ευρωπαϊκή δημοκρατία. Θα πρέπει να καταδικάσουμε κάθε μορφή βασανιστηρίου, την κακοποίηση εκρατουμένων σε οποιοδήποτε συνθήκες, ακόμη και όταν μιλάμε για, την, για τον αγώνα κατά της θερμοκρατίας. Δεν μπορεί η ανθρώπινη ζωή να θεωρείται ένα σημείο για ε, να το εξαφανίσει κανείς ή μια υπαρξιακή στατιστική. Ευχαριστούμε κύριε Καπούτο. Ο κύριος Καρίνς από το ΕΛΚ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πριν από λίγες εβδομάδες ο Πάπας βρισκόταν σε αυτή την αίθουσα και μας είπε ότι Ευρώπη, αν δεν παραμείνει σταθερή στις αξίες της, θα χάσει τη ρότα της, την πορεία της. Εδώ λοιπόν μιλάμε για ε, αγώνα κατά της θερμοκρατίας. Όμως κάποιοι επιβιώσαμε από τις επιθέσεις των Ταλιμπάν και από άλλους εξτρεμιστές. Αυτοί που μας επιτίθενται, επιτίθενται διότι θέλουν να μας αποσπάσουν τις αξίες μας. Αυτό θέλουν να μας πάρουν. Μην τους επιτρέψουν να το κάνουν, να το με τις αντιδράσεις μας θα έπρεπε να του δείξουμε με τις δράσεις μας ότι προσπιζόμαστε τις αξίες μας. Δεν επικρίνω μόνο τις ΗΠΑ, αλλά όσους σιωπηροί παρέμειναν μάρτυρες αυτά τα γεγονότα, ε, ε, συμπεριλαμβανομένων μερικών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Κάποιοι διευκόλυναν αυτές τις παράνομες ενέργειες σε κάθε περίπτωση. Σήμερα δεν έχουμε καμία εγγύηση για κανέναν από τους πολίτες μας ότι δεν θα μπορούσε να πέσει θύμα τέτοιων ενεργειών. Και οι κυβερνήσει μας ακόμη αποκρύπτουν στοιχεία και γεγονότα. Έχουμε μια επιλογή, συνάδελφοι. Είτε θα ενωθούμε και θα προσπίσουμε τις αξίες μας, είτε θα διαιρεθούμε και θα χρειαστεί να υποστούμε τις συνέπειες. Ευχαριστώ. Uh, thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, ο Γιώζου Ράντος από την ε, ομάδα των φιλελευθέρων και δημοκρατών. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι η η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο έχουν λάβει σαφή θέση όσον αφορά το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των ε, δικαιωμάτων του ανθρώπου και των ε, δημοκρατικών αξιών γενικότερα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που όλοι ε, σχεδόν ομόφωνα έχουμε λάβει μια άποψη αρχής παρά κάποιες παραφωνίες. Ωστόσο υπάρχουν κράτη-μέλη, συγγνώμη, υπάρχουν κράτη ε, μερικά ε, των οποίων είναι και στον δυτικό ανεπτυγμένο κόσμο, όπου όλα αυτά που λέμε δεν είναι τόσο προφανή. Δηλαδή, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όταν ε, μπαίνει στην πλάστικα μαζί με την ασφάλεια, δεν θα πρέπει να υπολείπεται. Αυτό που έκανε ο κύριος Ομπάμα, όπως ξέρετε, καταγγέλλεται από ορισμένου ε, γερουσιαστέ των ΗΠΑ που καταγγέλουν ε, τι παραβιάσει αυτέ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει οπωσδήποτε να χαιρετήσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει και ο πρόεδρο. Και τώρα ο κύριο Χουαρίστη για ένα λεπτό, παρακαλώ. Πρόεδρε, μιλάμε για την χρήση βασανιστήριων από πλευρά τη CIA. Τι γίνεται όμω με τι χώρε μέλη είναι συνένοχοι. Εφόσον υπήρξαν στην Ευρώπη κέντρα κράτησης τέτοιων ε, ανθρώπων που βασανίστηκαν. Κύριε Επίτροπε, υπογραμμίσαμε πριν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να καταπολεμήσει τη χρήση βασανιστερίων τόσο στην Ευρώπη όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Είπατε ότι πρέπει να διωχθούν οι υπεύθυνοι. Τι γίνεται με τις Ηνωμένε Πολιτείε όπου υπάρχει ατιμορρησία. Εδώ στην Ευρώπη, στη Μαδρίτη, έχουμε 28 Βάσκους οι οποίοι διώκονται, γίνεται δίκη τους αυτή την εποχή και βάσει βάση του πρωτοκόλου της ε, Κωνσταντινούπολης βλέπουμε ότι και αυτοί εμπλέκονται σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα βασανιστήρια. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να ερευνούνται περισσότερο και τέτοιες περιπτώσεις βασανιστήριων που έχουν γίνει και σε Βάσκους ή Καταλάνους κρατούμενους. λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, από το Γενάρη του 2002 δώσαμε ε, την ε, δυνατότητα στους, στις ΗΠΑ να συγκεντρώσουν 200 υπόπτους για τρομοκρατία, οι οποίοι περίμεναν επιμήνες ε, απομονωμένοι και κρατούμενοι ε, και επί 13 χρόνια ακολούθησαν καταγγελίες, εκατοντάδες καταγγελίες δημοσιογράφων και μη κυβερνητικών οργανώσεων για τις μυστικές φυλακές της ΗΠΑ και ανά τον κόσμο. Ακόμη και το Ευρωκοινοβούλιο συζήτησε ξανά και ξανά το θέμα και εξέφρασε τις ανησυχίες του με διάφορα ψηφίσματα. Όμως κάποια κάτι μέλη φαίνεται ότι κυριολεκτικά συνεργάζονταν με την CIA και προχωρούσαν σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριος Ομπάμα στην προεκλογική του εκστρατεία είχε τοποθετηθεί κατά του Γκαντάναμο και των πρακτικών τη. Όμως τελικά φαίνεται ότι αμβλήθηκε και η δική του βούληση να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδικάσει τα αφρικαλαία βασανιστήρια που διαπραχθήκαν με την Αμερικανική κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τώρα ο Επίτροπος ε, κ. Αβραμόπουλος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση σε αυτό το χώρο για την ε, έκθεση της Γερουσίας έφαρε μαζί με τα στοιχεία που μας δίνει η έκθεση στην επιφάνεια μια σκληρή πραγματικότητα μια σκληρή αλήθεια και θέτει όλους μας πραγματικά πρώτων ευθυνών μας και αξίζει αυτήν την έκθεση να τη χαιρετήσουμε. διαπιστώνω ότι όλες οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου σε αυτό το χώρο καταδικάζουν απερίφραστα τα βασανιστήρια και κάθε πρακτική που κινείται έξω από τα όρια του κράτους δικαίου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των αρχών και των αξιών πάνω στις οποίες έχει θεμελιωθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. είπα στην εισήγησή μου ότι τα βασανιστήρια είναι ένα έγκλημα και όσοι είναι υπόλογοι είναι ευθύνη των ιδίων των κρατών να τους τιμωρούν. ακούστηκε όμως και μια κριτική σε αυτό το χώρο ότι η ευρώπη δεν μάλλον σε πολλές περιπτώσεις ανέχθηκε. θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ευρώπη δεν ενέκρινε ποτέ αυτές τις πρακτικές που προσβάλλουν την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. μάλιστα για το λίγο χρονικό διάστημα που βρίσκομαι και εγώ κοντά σα εκείνο που καθημερινά βλέπω μπροστά μου είναι η υποχρέωσή μα να τα προστατεύουμε. οι εργασίε αυτή τη σημερινή εδώ συνέλευση όπω και η έρευνα τη επιτροπή τη γερουσία των ηνωμένων πολιτειών καταδεικνύουν τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει ο δημοκρατικός έλεγχος η δημοκρατική εποπτεία όσον αφορά στην εθνική ασφάλεια και την επιβολή του νόμου. οι πρακτικές που ανεδείχθησαν μέσα στη συζήτηση και που συζητήσαμε σήμερα εδώ δείχνουν ότι η προάσπιση και η πρόθεση των θεμελιωδών δικαιωμάτων απαιτούν συνεχείς προσπάθειες και επαγρύπνηση και ναι θα συμφωνήσω μαζί σας ότι την ευθύνη τη μοιραζόμαστε όλοι και τα κράτη μέλη. Και είμαι βέβαιος ότι ο Προεδρεύων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που βρίσκεται σήμερα εδώ θα μεταφέρει τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη. Θυμίζω όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ακούστηκαν και κάποιοι αφορισμοί ότι η έρευνα της επιτροπής της γερουσίας των ηνωμένων πολιτειών της αμερικής είναι αποτέλεσμα δημοκρατικού και κοινοβουλευτικού ελέγχου. το καλωσορίζουμε ως μια όριμη αντίδραση μιας δημοκρατικής κοινωνίας και θυμίζουμε ότι η δημοκρατία έχει τους θεσμούς έχει τη δύναμη και την θέληση να προστατεύει τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του. Φτάσαμε στο σημείο αυτό να κάνω μια αναφορά σε κάτι σημαντικό κατά τη γνώμη μου που είπε ο πρόεδρος ομπάμα ο οποίος όπως γνωρίζετε απαγόρεσε τα βασανιστήρια όταν ανέλαβε πρόεδρος. I quote, Today's report can help us η σημερινή έκθεση μπορεί να μας επιτρέψει να αφήσουμε αυτές τις τεχνικές εκεί που τους αρμόζει στο παρελθόν. Κάποιοι εκ των βουλευτών αναφέρθηκαν στον Κουαντάναμο. Τη θέση της Επιτροπής την ακούσατε στην αρχή και την επαναλαμβάνω. Και η θέση μας είναι σαφής και συνεπής. Ναι, ζητούμε το κλείσιμο του Κουαντάναμο. Τη στάση αυτή την έχουμε τηρήσει, κυρίες και κύριοι βουλευτές, με συνέπεια όσον αφορά όχι μονάχα στην επαόριστον κράτηση υπόπτων τρομοκρατίας στον γκουαντάναμο αλλά στη θανατική ποινή σας θυμίζω στη φυλάκιση ανηλίκων και άλλα σημαντικά ζητήματα που άπτονται των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. έγινε αναφορά και στην αντιτρομοκρατική συνεργασία ανάμεσα στην ευρωπαϊκή ένωση και τις ηνωμένες πολιτείες της η συνεργασία αυτή είναι πολύ σημαντική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την προστασία των λαών μας. σε επίπεδο ευρωπαϊκής ένωσης έχουμε συνάψει συμφωνίες με τις ηνωμένες πολιτείες αμερικής για σειρά πρωτοβουλειών που διευκολύνουν τη συνεργασία αυτή και την καθιστούν περισσότερο αποτελεσματική και σύμφωνη πάντα με τα θεμελιώδη δικαιώματα. η ευρωπαϊκή ένωση και τα κράτη μέλη της καθώς και οι ηνωμένες πολιτείες της αμερικής έχουν την κοινή ευθύνη να διασφαλίζουν ότι η αντιτρομοκρατική συνεργασία τους σέβεται απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου και κατά περίπτωση το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το δίκαιο περί προσφύγων. εμείς και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό θα συνεχίσουμε να θέτουμε και να συζητάμε τα θέματα αυτά με τις ηνωμένες πολιτείες αμερικής και να εκφράζουμε όπου χρειάζεται τις ανησυχίες μας και τους προβληματισμούς μας αλλά και τις προτάσεις μας για καταστάσεις που είναι αντίθετες προς τις αξίες και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ευρωπαϊκή ένωση στις ίδιες αξίες και αρχές που στηρίζεται το αμερικανικό δημοκρατικό οικοδόμημα. η ιδιαίτερη προσοχή που δίνει το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στα εν λόγω θέματα μας παρέχει πολιτική στήριξη και δημοκρατικό έλεγχο για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι ανησυχίες θα αντιμετωπίζονται με τρόπο ισορροπημένο και σωστό ενώ ταυτόχρονα δεν μας επιτρέπει να επαναπαυόμαστε. το βασικό συμπέρασμα από τη συζήτηση αυτή σήμερα είναι ότι η ευρωπαϊκή ένωση και οι δημοκρατικοί της θεσμοί είναι οι θεματοφύλακες των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δημοκρατικών μας κατακτήσεων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Και τώρα θα ζητήσω από τον κύριο Ντελαβέντοβα να μιλήσει εκ μέρους του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ για αυτήν την έντιμη ανταλλαγή απόψεων που ήταν και πλούσια, όπως είπατε. Πρέπει να, να βεβαιωθούμε ότι οι παραβιάσεις για τις οποίες έγινε λόγο στην έκθεση της Αμερικανικής Γερουσίας και που συζητήσαμε σήμερα δεν θα επαναληφθούν με πρόσχημα την ε, καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Πρέπει να γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Ευρωκοινοβούλιο έχει σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει στον διάλογο, τον διατλαντικό διάλογο για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και το ανθρώπινο, ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώ και το ανθρωπιστικό δίκαιο. Ξέρετε ότι μπορείτε για την πολιτική κατά της τρομοκρατίας να εκφράσετε τις απόψεις σας απευθείας του συναδέλφου σας το, της ε, Αμερικανικής Γερουσίας. Και είδαμε πώς οι ανησυχίες μας μπορεί να επηρεάσουν την Αμερικανική πολιτική. Αυτή τη στιγμή στο Κογκρέσο συζητάτε το θέμα της παρακολούθησης και προστασίας δεδομένων καθώς και ο σεβασμός του ιδιωτικού βίου. Το Κογκρέσο καταψήφισε ένα νομοσχέδιο που ε, συμπεριλάμβανε ένα πρόγραμμα μεγάλο ενδιαφέροντας για τους Αμερικανούς, οπότε σημαντικό θα είναι και το Ευρωκοινοβούλιο να τοποθετηθεί ως προς την σκοπιά που έχουν θετήσει οι γερουσιαστές των Ηνωμένων Πολιτειών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ιδιωτικό βίο. Θα, ε, θα πρέπει επίσης να ε, βεβαιωθούμε ότι συνεχίζονται και μεταρρυθμίσεις και σε άλλες περιοχές του κόσμου, που ε, στις περιοχές της, Βορείου, της χώρας της Βορείου Αφρικής, ώστε να υπάρχει ένας πραγματικός έλεγχος, όπως υπόθηκε, δημοκρατικός έλεγχος, όπως υπόθηκε αρχικά η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ σε θέματα καταπολέμησης Μοκατίας παραμένει θεμελιώδης σημασίας. Ο Ευρωκοινοβούλιο έχει εδώ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει σε ό,τι αφορά τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, αλλά και το Terrorist Finance Tracking Program ή το Μητρό των Ονομάτων Επιβατών για την ε, μετακίνηση επιβατών μεταξύ ε, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πρέπει να δούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τον ιδιωτικό βίο ακόμα και με την περίπτωση του ασφαλού λιμένα. Θα πρέπει λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Πολιτείε να δεχτούν την κοινή τρομοκρατική απειλή που αντιμετωπίζουν, ε, όπω από το Ισλαμιστικό κράτο ε, και του αγωνιστέ του, και θα πρέπει με τα προηγμένα εργαλεία που διαθέτουμε ή την ανταλλαγή δεδομένων να φροντίσουμε την απειλή αυτή να την αναχαιτήσουμε, αλλά με το σωστό τρόπο που θα ε, επιτρέπει και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είμαι πεπισμένο ότι η συζήτηση αυτή για την τρομοκρατία σε συνδυασμό όμω με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συνεχιστεί και στι δύο όχθε του Ατλαντικού και σε αυτό το Ευρωκοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Eh, Ευχαριστούμε τον Υπουργό. Και τώρα Εάν θέλετε να πάρετε το λόγο με κίτρινη κάρτα, δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη φάση τη διαδικασία. Ή δεν μπορείτε να απευθυνθείτε στην Επιτροπή ή στο Συμβούλιο με αυτήν την μορφή. Διαδικαστικό. Θα ήθελα το Συμβούλιο να κάνει δήλωση για το θέμα που συζητάμε εδώ σήμερα το απόγευμα. Εγώ διαπίστωσα ότι το Συμβουλίο ούτε στην εισαγωγή του ούτε στα συμπεράσματα είπε κάτι για τον ρόλο. Δεν έγινε καμία δήλωση από το Συμβούλιο όταν συζήτησαν την ε, στρατηγική. Δεν είπε τίποτα. Για μένα το Συμβούλιο δεν έκανε καμία δήλωση, δεν απάντησε. Σας ευχαριστούμε. Αυτή είναι η προσωπική σας άποψη. Την εκφράσατε δημοσίως. Το Συμβούλιο μας αποσωπείται εδώ. Ολοκληρώνεται η συζήτηση.